Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε την ημέρα μας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ας ε, ξεκινήσουμε αμέσως με την ακρόαση της Επιτρόπου που είναι αρμόδια για τις ε, μεταφορές και τις μελλοντικές προοπτικές στην πολιτική μεταφορών. Καλώς ήρθατε κυρία Βαλεάν, στην Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ απλό το πλαίσιο. Η κυρία Βαλεάν θα πάρει το λόγο για 10 λεπτά για να μας παρουσιάσει το όραμά τη ε, για τη θητεία αυτή. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στους συντονιστές. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Βαλεάν για να απαντήσει και κατόπιν θα έχουμε και ένα δεύτερο γύρο συζητήσεων για όσους θέλουν να τοποθετηθούν. Καλώς ήρθατε. Έχουμε βεβαρημένη ημερησία διάταξη μεταξύ της Πράσινης Συμφωνίας ε, και όλα όσα έχουμε τελειώσει με την προηγούμενη θητεία και των ε, προκλήσεων. Καλώς ήρθατε κύριε Βαλεάν. Έχετε το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που λέω ότι είναι γεμάτη η ημερήσια διάταξή μας ε, με πολλά θέματα και σίγουρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ζωή μας για το επόμενο χρονικό διάστημα. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί πρώην συνάδελφοι, χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας ενημερώσω για το που βρισκόμαστε με τους συνεχιζόμενους φακέλους για τις μεταφορές ε, και να σας παρουσιάσω τις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της Κομισιόν στον τομέα των μεταφορών. Γνωρίζετε ότι θέλω να συνεργαστώ μαζί σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ιδίω με την Επιτροπή σας. Νομίζω ότι από κοινού μπορούμε να οικοδομήσουμε ευφύ συστήματα μεταφορών και βιώσιμα που αξίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ ταυτόχρονα θα διατηρήσουμε προσιτή, διαθέσιμη και ασφαλή κινητικότητα για όλους. Αυτή είναι η υπαριθμόν ερωτητά μου που θα καθοδηγήσει το πολιτικό μου θεματολόγιο την επόμενη πεντετία. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία έχει στόχο να καταστήσει την ευρωπαϊκή οικονομία προς προ εκπομπέ το 2050 και φυσικά οι μεταφορέ θα έχουν ρόλο κλειδί. Επίση, οι μεταφορέ είναι πολύ σημαντικέ για την ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή οικονομία. Προκειμένου η βιομηχανία τη Ευρώπη να μην είναι ανταγωνιστική, θα πρέπει να εξυπηρετείται από ε, ένα ε, σύστημα μεταφορών και μελετίας ε, που θα λειτουργεί στην εντέλεια. Πριν να στραφώ σε συγκεκριμένα ζητήματα, να πω δύο λόγια για την οδική ασφάλεια. Μόλις ήρθα από τη Στοκχόλμη, όπου περιβρεθεί στην Παγκόσμια Υπουργική Διάσκεψη ε, για την οδική ασφάλεια και με εντυπωσίασε η παρουσία των Υπουργών και όλοι συμφώνησαν ε, ότι είναι πραγματικά απαράδεκτο ε, το κόστος του 1,35 σε εκατομμυρίων από τα δικά ατυχήματα. Ε, και είπαμε ότι καταρχήν χρειαζόμαστε μείωση ε, κατά 50% του στόχου της θνησιμότητας. Αυτός είναι ο παγκόσμιος στόχος και θα συνεργαστούμε με τα Ηνωμένα Έθνη για να πετύχουμε αυτό το στόχο παγκοσμίω. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να συνεχίσει να δείχνει η ηγετική θέση ισχυρή σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώ θα προωθούμε για ένα πιο ασφαλή κόσμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη έχει δεσμευτεί να βλάβει μέτρα οδική ασφάλεια για να μειώσει ε, τα ατυχήματα στο δρόμο, τα θανατηφόρα αλλά και του τραυματίε κατά 50% και θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πετύχει ε, το φιλόδοξο στόχο μέχρι το 2050 να μην έχουμε ε, καθόλου θνησιμότητα στο δρόμο. Τώρα θα έρθω στην ευφυή κινητικότητα και στη βιώσιμη στρατηγική. Η στρατηγική αυτή θα είναι η πρωτοβουλία Ναυαρχίδα για το 2020 για τις μεταφορές. Θα δούμε πώς μπορούν να συνεισφέρουν οι μεταφορές στην ουδετερότητα μέχρι το 2050 και πώς χρησιμοποιούμε τις ψηφιακές τεχνολογίες στον τομέα μας. Η στρατηγική θα περιγράφει τα κύρια μέτρα που θα ληφθούν στις μεταφορές, όπου η Κομισιόν θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξουν δράσεις πολιτικής τα επόμενα έτη. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει φιλόδοξα μέτρα για τη μείωση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα κατά 90% μέχρι, 50, ε, μέχρι το 2050 και την μείωση τη ρήπανση σε όλου του τρόπου μεταφορά. Επίση, θα δούμε πώ θα εκμεταλλευτούμε την ψηφιοποίηση και την αυτοματοποίηση και θα προωθήσουμε την συνδεσιμότητα στο επόμενο επίπεδο. Θα εξετάσει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα, πώ να αντιμετωπίσει τι κοινωνικέ προκλήσει και πώ θα διατηρήσει διαθέσιμη προσιτή και ασφαλή κινητικότητα σε όλου και στι απομακρυσμένε περιοχέ να τονίσω τις, ε, τους κύριους τομείς δράσης στρατηγικής σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Καταρχήν, η στρατηγική στοχεύει στο να προωθήσει ε, την ε, υιοθέτηση καθαρών οχημάτων και εναλλακτικών καυσίμων ε, για τις οδικές θαλάσσιες ε, και αεροπορικές μεταφορές. Ε, θα πρέπει να επιταχύνουμε την ανάπτυξη και την ετοιμότητα των αγορών για τις νέες τεχνολογίες και να έχουμε ανάπτυξη υποδομών και παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων. Θα πρέπει να είμαστε ταχείς με συγκεκριμένες δράσεις για φέτος θέτω δύο προτάσει στο πρόγραμμα εργασία τη Κομισιόν. Καταρχήν, εναλλακτικά βιώσιμα καύσιμα για την αεροπλοεία και μία για τι θαλασσίε μεταφορέ. Επίση, θα έχουμε μια πρόσκληση χρηματοδότησης για να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη ε, δημοσίων τόπων για τον ανεφοδιασμό ως μέρος της στρατηγικής της υποδομής για τα ελεκτικά καύσιμα. Επίσης, ε, η αναθεώρηση του κανονισμού TNT των διαδικτύων ε, ΔΕΔ μεταφορών προβλέπεται για το 2021 πρέπει να αυξήσουμε ε, την αποτελεσματικότητα σε όλο το σύστημα και θα εργαστούμε για μια νέα πρόταση για ολιστική προσέγγιση για να πρασινίσουμε τις μεταφορές εμπορευμάτων στην Ευρώπη και αναμένεται να σας παρουσιάσω συγκεκριμένες προτάσεις μέχρι το 2021, το 2021. Οι σιδηροδρομικέ μεταφορές είναι σημαντικές ε, για τη μείωση των εκπομπών. Ε, όχι μόνο μπορεί να μας βοηθήσει να απανθρακοποιήσουμε τις μεταφορές, αλλά μας βοηθάει και να μειώσουμε και την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αξιολογούμε τον κανονισμό για τους ε, διαδρόμους, για τις εμπορικές δρόμικε μεταφορέ, καθώ θα πρέπει να προωθήσουμε ε, ουσιαστικά αυτό τον κλάδο συνεισφέροντα και στου στόχους τη συμφωνία Επίση, ξέρετε ε, για το συνδυασμένη οδηγία μεταφορών, ξέρετε ότι έχουμε προτείνει να αποσύρουμε την πρότασή μα γιατί δεν ήταν πλέον αρκετά φιλόδοξα τα κείμενα που συζητήθηκαν στο Συμβούλιο. Επίσης, ε, θέλουμε να αυξήσουμε και να διαχειριστούμε καλύτερα την ε, ικανότητα ε, των οδών εσωτερική συναυσιπλοείας. Επίσης, σε με το Green Deal έχουμε και τρίτο τομέα κλειδί. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουν επιλογέ οι καταναλωτέ ό,τι αφορά του τρόπου μεταφορά ε, και τα μοντέλα ε, κινητικότητα χαμηλών εκπομπών. Η στρατηγική θα περιγράφει πώ μπορούμε να συντορικοποιήσουμε το εξωτερικό κόστο των μεταφορών μέσω τη τιμολόγηση, ώστε θα διατηρήσουμε την προσβασιμότητα ε, και φτηνέ μεταφορέ. Επίση, θα ήθελα να εξετάσουμε και μέτρα για το πώς μπορούμε να ενημερώσουμε τους ε, ε, καταναλωτές για εναλλακτικέ ε, μεταφορές. Η τέταρτη, ο τέταρτος κλάδος εργασίας σε σχέση με την πράσινη στρατηγική πρέπει να αυξήσουμε τις επενδύσεις για λύσεις χαμηλών εκπομπών και τις υποδομές. Θα έχουμε ειδική χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σίγουρα δεν αρκεί η στρατηγική. Θέλει να διασφαλίσει καλύτερο συντονισμό των διάφορων μέσων χρηματοδότησης, καθώς και να κινητοποιήσει καλύτερη ιδιωτική χρηματοδότηση χρηματοδότηση. Τώρα θα αναφερθώ σύντομα σε ένα άλλο στοιχείο που συνδέεται συχνά με τη μελλοντική στρατηγική, να είναι πιο ευφυέ το σύστημα μεταφορών. Η ψηφιοποίηση και η καινοτομία είναι βασικέ για να αυξήσουμε την αποδοτικότητα των συστήματων μεταφορών. Η ψηφιοποίηση είναι καλά νέα για το περιβάλλον, αλλά και για την προσβασιμότητα και την ασφάλεια. Και θα διασφαλίσουμε ότι επίση είναι καλά νέα για τι επιχειρήσει και του πολίτε. Για να ελοπιθεί αυτό θα πρέπει να θέσουμε τι κατάλληλε συνθήκε. Ε, τα δεδομένα είναι το κατέργαστο υλικό τη ψηφιοποίηση και όπω θα έχετε δει στη στρατηγική για τα δεδομένα που δημοσιεύτηκε χθε, θα εργαστούμε σε ένα κοινό ευρωπαϊκό χώρο κινητικότητα δεδομένων ε, προκειμένου να αναπτύξουμε ένα ευφυέ σύστημα μεταφορών. Το σύστημα που έχουμε είναι όλο ένα και πιο συνδεδεμένο και στο εγγύς ε, μέλλον θα είναι όλο ένα και πιο ε, αυτοματοποιημένα και αυτόνομο οχήματα που θα κουβαλούν τους επιβάτες και τα αγαθά. Προκειμένου η Ευρώπη να παραμείνει σε ηγετική θέση θα πρέπει να επικεντρωθούμε όχι μόνο σε καινοτόμε τεχνολογίε, αλλά και να διασφαλίσουμε την αποδοχή από την κοινωνία. Οι λαοί τη Ευρώπη θα πρέπει να μα υποστηρίξουν αν θέλουμε να αναπτύξουμε γρήγορα νέε τεχνολογίε και να εκμεταλλευτούμε τα μάλλα τι νέε ευκαιρίε. Ενώ το θέμα της αηφορίας και της ευφυΐας ε, σίγουρα θα καθορίσουν τις θεματικές μας, ε, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είναι ανταγωνιστικές οι μεταφορές θα πρέπει να δούμε όλες ε, τις προκλήσεις και τα συνάφη μέτρα ως ευκαιρία για να ε, μεταμορφώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ε, μια ευημερούσα κοινωνία με μια μοντέρνα και ανταγωνιστική οικονομία. Ένα λεπτό μου μένει. Αν θέλετε μπορώ να μπω στο πρόγραμμα εργασίας. Συγγνώμη, είχαμε πολλά στοιχεία να φέρουμε στην αρχή. Λοιπόν, για το πρόγραμμα εργασία για το 2020 θα επικαιροποιήσουμε την οδηγία για την άδεια οδήγηση για να αντικατοπτρίσουμε τι κοινωνικέ αλλαγέ και τον αντίκτυπο τη τεχνολογία ε, αρρωγή στην οδήγηση. Ε, Επίση, ε, παρακολουθούμε την αναθεώρηση τη οδηγία για τα εφή συστήματα μεταφορών και την κατοξιδότηση πράξη CITS. Έχουμε 17 κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν μια ευρυδική στρατηγική. Η θέλει να δώσει ασφάλεια δικαίου στου επενδυτέ και στους όσου ε, υιοθετήσουν έγκαιρα, προκειμένου να υπάρχει ασφαλεία και εμπιστοσύνη. Επίση, πιστεύω ότι θα υπάρχει πρόοδο ε, σε έναν αριθμό φακέλων τη αεροπορία. Ξέρετε, γιατί πρέπει να ο κανονισμό για τα σλότ. Είναι σημαντικό φάκελο που θα μα βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τη συμφόρηση στα αεροδρόμια της Ευρώπης, οι νέες πρωτοβουλίες θα εξετάσουν την ανάγκη να θεωρηθούν οι κανόνες για τους φόρους των εδρομών και για τις ανερίες υπηρεσίες, γιατί αυτά έχουν μεγάλο αντίκτυπο ε, και στο κοινό και στους εργαζομένους ε, και στον κλάδο. Για τον Brexit θα περιορίσω τα σχόλιά μου τώρα, απλώς θα πω ότι δεσμευόμαστε να διατηρήσουμε τους δεσμούς μεταφορών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, ώστε να ήταν περισσότερο στο μέλλον, καθώς θα προσδιορίζουμε τις ε, νέες σχέσεις. Δεν θα είναι εύκολες οι διαπραγματεύσεις, αλλά θα αναφερθώ σε αυτό το θέμα αργότερα αργότερα, αν θέλετε, να το δούμε ξεχωριστά. Θα σταματήσω εδώ και μάλλον θα αναφερθώ και σε άλλα θέματα, ανάλογα με τις ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε, κυρία Επίτροπε. Και χωρίς άλλη χρονοτριβή, περνάμε στους συντονιστές. Για τρία λεπτά ο καθένας. Πρώτα, κυρία Μπάρμπαρα Δελόρ. Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την Επίτροπο για την παρουσίαση της στρατηγικής. Ε, Αναφέρατε τις ε, πράσινες εμπορευματικές μεταφορές και σίγουρα οι σιδηρόδρομοι θα παίξουν κέριο ρόλο σε αυτή την προσπάθεια για μια πιο φιλοπεριβαλλοντική πολιτική μεταφορών. Σίγουρα οι σιδηρόδρομοι θα αποτελέσουν τη λύση κλειδί για τις περισσότερες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στις μεταφορές. Δυστυχώς όμως ο σιδηροδρομικός κλάδος πόρο απέχει από την αξιοποίηση στο έπακρο του δυναμικού του δεδομένης της ε, συνεχούς αυτοματοποίησης της οδικές μεταφορές, το μέλλον και τα επόμενα μέσα χρόνια θα είναι κρίσιμα για το μέλλον και των σιδηρομεταφορών, σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρώπη. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να καταργήσουμε τους γραφειοκρατικούς και προστατευτικούς κανόνες που παρεμποδίζουν το γνήσιο και θεμητό ανταγωνισμό και στις ε, σιδηροδρομικές μεταφορές. Εσείς τι μέτρα σκοπεύετε να υιοθετήσετε για να στηρίξετε τις σιδηροδρομικές μεταφορές και να γίνουν ουσιαστική εναλλακτική λύση ω προς τις οδικέ μεταφορές. Σας διαβεβαιώ για την αμέριστη υποστήριξη τη Επιτροπής Μεταφορών στο στόχο μας. Και θα περάσω στα γερμανικά που είναι η μετρική μου γλώσσα για το δεύτερο θέμα που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Κύριε Επίτροπε, την προηγούμενη εβδομάδα όταν επισκεφθήκατε το Τυρόλο αναφέρατε ότι ο διάδρομος Μπρένερ δεν ανήκει στους Τυρολέζους αλλά σε όλους τους Ευρωπαίους και πράγματι έχετε δίκιο. Είναι όμως ο ζωτικός μας χώρος και γι' αυτό πρέπει να τον προστατεύσουμε. Αν ένας διάδρομος ανήκει σε όλους τους Ευρωπαίους τότε αυτό ισχύει και στους δρόμους που οδηγούν προς το διάδρομο. Και γιατί ε, πρέπει να περιμένουμε και να βλέπουμε ότι δεν γίνονται τα απαραίτητα έργα. Εάν τα μέτρα για το Τυρόλο τα χαρακτηρίζεται μονομερή μέτρα, τότε και εγώ πρέπει να πω ότι το ότι δεν κατασκευάζονται δρόμοι που οδηγούν στο διάδρομο και αυτό είναι ένα μονομερές μέτρο. Τι προτίθεται λοιπόν να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξευρεθεί μακροχρόνια λύση, πρέπει να ληφθούν μέτρα. Το πρόβλημα του Μπρένερου είναι ε, ένα πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να συμπεριληφθεί και η Ελβετία στη λύση του προβλήματος. Τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε η ε, <clears throat> διέλευση μέσω Ελβετίας να περιστεί και έτσι ώστε να επωφεληθούν όλοι με το περίφημο πρόγραμμα Single European Sky το Τυρόλο έχει κάνει ό,τι μπορούσε να κάνει και πρέπει να λάβει μέτρα για να προσφέρει οδική ασφάλεια. Από το 2013 μέχρι το 2018 οι οδικές μεταφορές αυξήθηκαν κατά 43%. Εσείς λοιπόν τι προτίθεστε να κάνετε έτσι ώστε οι στόχοι της Λευκής Βίβλου που προβλέπουν μείωση κατά 50% να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί. Κύριε Επίτροπε, πρέπει να σας πω ότι εξεπλάγει που την προηγούμενη Παρασκευή είπατε ότι το Τυρόλο θα πρέπει να αποσύρει τα μέτρα. Αλλά εγώ θέλω να στρέψω το βλέμμα στο μέλλον. Εμείς οι Τυρολέζοι είμαστε πεπισμένοι Ευρωπαίοι και έτσι θέλουμε τα προβλήματα να λύνονται από κοινού. Ε, το πρόβλημα της, ε, των μεταφορών και της οδικής ασφάλεια δεν μπορεί να το επομίζεται μόνο το Τυρόλο. Ευχαριστούμε κυρία Τάλερα, αλλά παρακαλώ να εμένετε στο τρίλεπτο συντονιστέ. από σεβασμό προς τους ακόλουθους ομιλητές κύριος Ντάνιλσον. Σας ευχαριστώ. Και ευχαριστώ και την Επίτροπο Βαλεάν που ήρθε σήμερα στην Επιτροπή μας και την ευχαριστώ που την περασμένη εβδομάδα ήταν στο Στρασβούργο και συζητήσαμε πολύ σημαντικά θέματα οδικής ασφάλειας. Οι μεταφορές, όπως είπατε και εσείς, θα είναι ε, σημαντικός παράγοντος ε, που θα μας βοηθήσει να υλοποιήσουμε το στόχο μας για την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Περιμένουμε λοιπόν τη στρατηγική σας ε, στη συνέχεια του χρόνου και χαίρομαι που ήδη από φέτος θα προταθεί νομοθεσία για τα εναλλακτικά καύσιμα στην αεροπορία. Γιατί θα πρέπει να αναλάβουμε άμεση δράση για να προωθήσουμε τα εναλλακτικά καύσιμα και στην αεροπορία. Εγώ όμως θα επικεντρωθώ σε ένα άλλο θέμα. Την επικείμενη αναθεώρηση του κανονισμού για τις αεροπορικές ε, υπηρεσίες. Σίγουρα ε, η αναθεώρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη και κάποιες κοινωνικές πτυχές της αεροπορίας και εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά συνδικάτα εδώ και χρόνια μας ζητούν να εγκύψουμε στο θέμα αυτό. Και πιστεύω ότι θα, έχουμε, πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον δύο τεινά σε αυτή την αναθεώρηση για τις κοινωνικές πτυχές. Καταρχήν, σήμερα τα πληρώματα αεροπλάνων σε πολλές περιπτώσεις υπόκεινται στις κανόνες, στο εργατικό δίκαιο και στα κοινωνικά δικαιώματα της χώρας προέλευσης, ακόμη και αν η βάση ε, της δραστηριοποίησης είναι άλλη χώρα αυτή η πρακτική είναι απαράδεκτη κατά τη γνώμη μας. Θα πρέπει να καταργηθεί και να διευκρινίσουμε το ενωσιακό δίκαιο στα θέματα αυτά και ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο για τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Γιατί έχουμε ευρωπαϊκές δικαστικές αποθέσεις και την ευρωπαϊκή νομολογία που μερικές φορές αντιβαίνει στην εθνική νομολογία και την ερμηνεία που δίνουν τα εθνικά δικαστήρια. Επίση, για το wet αυτή είναι μια προσωρινή μέθοδος για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του οι αεροπορικές εταιρείε, αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως τρόπος παράκαμψης των συλλογικών συμφωνιών με εξωτερική ανάθεση των δραστηριοτήτων τους. Επίσης, θα ήθελα να παροτρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρακτικές όπως το pay to fly, δηλαδή καταβολή τελών προκειμένου να πετάξει ο πιλότος για να εξασκηθεί. Θα πρέπει τέτοια συστήματα να καταργηθούν στην αεροπορία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε Μπαουσά Δίας. Κυρία Επίτροπε, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας ξαναβλέπουμε στην Επιτροπή μας για να ακούσουμε τις προτάσεις σας, αλλά και να ακούσετε και εσείς τις ανησυχίες μας και τις απορίες μας. Όπως σας θυμάστε, στις 14 Νοεμβρίου του 2019 είχατε έρθει στην Επιτροπή μας για να Παρουσιάστε τις κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματός σας. Τότε είχαμε ακόμη το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Βρετανούς ε, Ευρωβουλευτές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δυστυχώς έχει συντελεστεί πια το Brexit και οι Βρετανοί δεν είναι πια μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ξεκινήσουν έντονες διαπραγματεύσεις σε πολλούς τομείς και φυσικά και στις μεταφορές. Αλλά και στις μεταφορές ε, συμπεριλαμβάνεται η αεροπορία. Οπότε θα πρέπει να έχουμε σκληρές διαπραγματεύσεις και το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι φιλόδοξο, ισορροπημένο και να λαμβάνει υπόψη και την αεροπορική κυκλοφορία, την εναέρια ασφάλεια και την, ε, τα δικαιώματα των ε, αεροπορικών εταιριών σε αυτόν τον κλάδο της αεροπορίας. Και όταν το Νοέμβριο είχατε ζητήσει την έγκρισή μας για να αναλάβετε τη, τα καθήκοντά σας. Μιλήσαμε ε, και για την περίπτωση του αεροδρομίου του Γιβραλτάρ. Ε, ξέρετε ότι η Ισπανία δεν αναγνωρίζει την επικυριαρχία του Ηνωμένου Βασιλείου στο βράχο του στο... στην περιοχή του Γιβραλτάρ. Είναι το, ότι αν λάβει χώρα το Brexit, μα είχατε πει τότε, εγώ θα είμαι ε, πίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια και το Brexit όμως έχει υλοποιηθεί. Και δεδομένου ότι τώρα θα ξεκινήσουμε τις έντονε διαπραγματεύσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου για όλους τους τομεί και άρα και για τις μεταφορές και την αεροπορία. Θα ήθελα να αναφερθώ στις ευρωπαϊκές αρμοδιότητες για το Γιβραλτάρ και να κάνω δύο ερωτήσεις. Τι προβλέπετε για τις διαπραγματεύσεις μιας συνολικής αεροπορικής συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο και τι στοιχεία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για να εξασφαλιστεί η εναέρια διασυνδεσιμότητα μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικά ως προς το Γιβραλτάρ. Εσείς θα αναγνωρίσετε την κοινή κυριαρχία του αεροδρομίου του Γιβραλτάρ στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Και επαναλαμβάνω τις ευχαριστίες μου για την παρουσία σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις που θα μου δώσετε. Σας ευχαριστώ κύριε Μπαουσαντίας. Ο κύριος Εντέρ. Ευχαριστώ. Εγώ θα μιλήσω γερμανικά. <coughs> Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, ως Αυστριακός ε, Ευρωβουλευτής ε, Κύριε Επίτροπε, εξακολουθώ να έχω την εντύπωση της επίσκεψης ε, που κάνατε την προηγούμενη εβδομάδα στο Τιρόλο. Η επίσκεψη αυτή, πρέπει να σας πω, προκάλεσε μέχρι και αγανάκτηση. Κυρίως αυτά τα οποία υποτίθεται ότι είπατε εκεί. Εγώ δεν ήμουν παρόν, αλλά φέρεστε ότι είπατε ορισμένα πράγματα. Και αυτά μεταφέρθηκαν σε εφημερίδες. Όσον αφορά λοιπόν τη διέλευση από τον Μπρένερο, ε, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Η προκάτοχος της Μπούλτς ε, τον Δεκέμβριο του 2018 ανακοίνωσε ότι ε, αυτός ο διάδρομος είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου είπαν ότι την προηγούμενη εβδομάδα εσείς στην Αυστρία είπατε επ' αυτού ότι αυτό δεν σας είναι σημαντικό και πριν η Αυστρία αρχίσει να μιλάει για κάτι τέτοιο τέτοιο ε, θα έπρεπε να αρθούν οι περιορισμοί ε, μέσα από το διάδρομο, κάτι το οποίο είναι παντελώς απαράδεκτο ως θέση στην Αυστρία. Και θέλω να επισημάνω ότι πέρυσι ε, στο Βερολίνο εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα 10 σημείων με βάση το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Γερμανία και η Ιταλία θα πιέσουν είτε να αυξηθούν τα διόδια, το ύψος των διοδίων, είτε να επιταχυνθούν οι δρόμοι που οδηγούν σε αυτό το διάδρομο, να επιταχυνθούν τα έργα. Η δική σας επίσκεψη στο Τυρόλο άφησε την ακριβώς αντίθετη εντύπωση και γι' αυτό λοιπόν σας ερωτώ ευθέως. Αυτά τα οποία αποφασίσαμε το 2018 και το 2019, από κοινού τα αποφασίσαμε ότι θέλουμε να περιορίσουμε τη διέλευση από το Μπρένερο και έτσι να είναι πιο ακριβή η διέλευση, ε, να υπάρχουν και δρόμοι που θα είναι ε, παρακαμπτήριες οδοί, ε, αυτά να τα χρηματοδοτήσουμε χρηματοδοτήσουμε με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα λοιπόν αυτά τα οποία είπατε κατ' ουσίαν στηρίζουν αυτά που έχουμε αποφασίσει ή ισχύουν αυτά που ε, μου είπαν ότι προέκυψε ως εντύπωση από την επίσκεψή σας ε, στο Τυρόλο. Απομακρύνεστε από την ε, πολιτική και από ό,τι φαίνεται, είπατε στο Μπρένερο, ότι αν δεν μας αρέσει, ε, και ας φύγουμε και από την κοινή αγορά. Ε, εσείς λοιπόν, τι ακριβώς κάνετε στηρίζεται αυτά τα οποία αποφασίστηκαν πέρυσι το 2018 σχετικά με το ύψος των τελών των διοδίων μέσα από τον Πρένερο και των παρακαμπτηρίων αδών. Ευχαριστώ κύριε Ντέρο, κύριε Σταλούντα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κόσμος εξελίσσεται ραγδαία και προσαρμόζεται στην ανάγκη της βιωσιμότητας. Και οι πολίτες μας αλλάζουν πολύ πιο γρήγορα από τις πολιτικές μας. Και γι' αυτό έχουμε ένα και μεγαλύτερο λαϊκό κίνημα ε, χιλιάδων ή εκατομμυρίων συμπολιτών που προτιμούν το τρένο για τις μεταφορές τους και τις θεωρούν πιο βιώσιμες τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Και μάλιστα στη Σουηδία έχουμε ε, την ομάδα του Facebook ε, που προάγει τις ε, διακοπές και τα ταξίδια με τρένο. Είναι το μεγαλύτερα, η μεγαλύτερη ομάδα του Facebook. Και μάλιστα μερικοί συμπολίτε μα ε, εκνευρίζονται που το πολιτικό σύστημα δεν διευκολύνει τι βιώσιμε μεταφορέ ή τις μεταφορές με σιδηρόδρομο. Σε ό,τι αφορά την έκδοση, διασυνοριακή έκδοση εισιτηρίων, σε μερικά κράτη-μέλη είναι πιο εύκολο να κάνουν κράτηση για να ταξιδέψουν από τη μία πόλη στην άλλη. Αν όμω έχουν διασυνοριακό ταξίδι μεγάλη απόσταση, είναι πολύ πιο δύσκολο να κάνουν κράτηση του εισιτηρίου. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα των επιβατών και στι διασυνοριακέ μεταφορέ. Και να είναι σίγουρος ότι ο πολίτης, ότι θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά του θα έχουμε τον τριμερή διάλογο τώρα για τα δικαιώματα των επιβατών στι ε, σιδηροδρομικές μεταφορέ. Αν δεν επιτύχουμε όμω αυτή τη διαδικασία, τι προτάσει θα υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξασφαλίσει την πιο εύκολη ε, κράτηση εισιτηρίων σιδηροδρομικών ε, για μεταφορές διασυνοριακής μακράς απόστασης. Επίσης, τα νυχτερινά δρομολόγια των τρένων, όλο και περισσότερες, επιχειρήσει. και επενδύουν σε νυχτερινά δρομολόγια, αλλά όχι όλες και όχι σε όλες τις χώρες μέλη. Τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να διευκολύνει τους παρόχους ε, να δρομολογήσουν τέτοια νυχτερινά δρομολόγια που να είναι ταυτόχρονα και επικερδή για να έχει νόημα η επένδυση και σε αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Νταλούντε. Ο κύριο Ζωτόφσκι. Καλημέρα σα Για τρία λεπτά έχετε και εσεί το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Επίτροπε, Χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω την ευκαιρία να σας υποβάλω την ερώτηση για το πακέτο κινητικότητας, που βέβαια είναι επιτεύγμα της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας. Και στην τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία, εμείς περισσότερο αγγίπτουμε στην Νέα Πράσινη Συμφωνία και την προστασία του περιβάλλοντος. Βέβαια, με την εφαρμογή των μέτρων του πακέτου κινητικότητας, ίσως έχουμε αύξηση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα έως και 30% έχουν επισημάνει τα κράτη-μέλη. Επίσης, ε, το καμποτάζ ή η υποχρέωση της επιστροφής άδειων φορτηγών ε, μετά την παράδοση, όλα αυτά θα οδηγήσουν σε αύξηση των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Το εξετάσατε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τη δική σας θέση τη γνωρίζουμε. Συζητήσατε όμως για αυτό το θέμα με τον κύριο Φραν Τίμερμαν στον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για την Νέα Πράσινη Συμφωνία και ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του συνόλου των επιτρόπων, δηλαδή του συλλογικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, για τη μελέτη αντικτύπου που υποσχεθήκατε. Πότε θα υποβληθεί αυτή. Επίσης, πολλά έχουμε Πήγε για την οδική ασφάλεια στο Στρασβούργο πρόσφατα. Ήσασταν και εσείς παρούσα και μας μιλήσατε για αυτό το θέμα. Είπατε ότι θέλουμε να μειώσουμε κατά το ίμιση τα θανατηφόρα τροχέα. Αλλά μιλάτε για μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ γνωρίζουμε ότι σε κάποιες χώρες μέλη τα τροχέα είναι ακόμη περισσότερα και τα στοιχεία πολύ πιο τρομακτικά από τις άλλες χώρες μέλη. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στις χώρες που έχουμε τα περισσότερα τροχιά, γιατί ο κοινοτικός μέσος όρος είναι μέσος όρος ακριβώς. Επίσης, μιλήσατε για την πρόθεση των εναλλακτικών καυσίμων στην αεροπορία. Θα πρέπει όμως ε, να γίνει παραγωγή πρώτα αυτών των καυσίμων. Θα πρέπει να τα παρασκευάσουμε και να δημιουργήσουμε και χώρους αποθήκευσής τους. Προβλέπετε λοιπόν ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των επενδύσεων στον τομέα των εναλλακτικών καυσίμων για να έχουμε και κατάλληλες εγκαταστάσεις και χώρους αποθήκευσης. Θέλουμε λοιπόν επενδύσεις για την παραγωγή και την αποθήκευση των εναλλακτικών καυσίμων εφόσον θέλουμε να τα προωθήσουμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Ζωτόφσκη. Κυρία Κουντουρά. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Βαλεάν, κυρία Επίτροπε, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Σωστά έχετε εντοπίσει ως βασικές αρχές της στρατηγικής σας ε, τη βιωσιμότητα, την ψηφιοποίηση αλλά και τη δικαιοσύνη, ώστε όπως είπατε να μην μείνει κανένας πίσω στην προσπάθεια μετάβασης. Θα ήθελα λοιπόν να σταθώ σήμερα στις ανάγκες των πιο ευάλωτων περιοχών, των περιφερειακών, των ισιωτικών περιοχών Συγγνώμη. Η ύπαρξη συνδεσιμότητας με αξιόπιστα οικονομικά προσιτά μέσα μαζικής μεταφοράς τόσο για τις τοπικές μεταφορές όσο και για τις συνδέσεις με τα αστικά, εθνικά και ευρωπαϊκά κέντρα είναι ζωτική σημασία για τις περιοχές αυτές τόσο για την οικονομική αλλά και τη δημογραφική τους επιβίωση, ειδικά στην περίπτωση των νησιών οι αεροπορικές μεταφορές για τη σύνδεση των περιφερειακών χωρών με το κέντρο της Ευρώπης είναι σήμερα μονόδρομος. Ποια εναλλακτική υπάρχει για να ταξιδέψει κανείς από τις Βρυξέλλες στην Αθήνα, στη Λισαβόνα, στο Δουβλίνο ή στα κράτη-μέλη Μάλτα, Κύπρο. Σε αντίθεση βέβαια με άλλες περιοχές της κεντρικής Ευρώπης όπως είναι το Παρίσι, η Φραγκφούρτη, το Βερολίνο όπου το τρένο αποτελεί μια εξαιρετική και βιώσιμη εναλλακτική. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να διαφοροποιήσετε τη στρατηγική σας για τις αεροπορικές μεταφορές, ώστε να μην πληγεί η συνδεσιμότητα της περιφέρειας, την οποία εσείς έχετε θέσει ως προτεραιότητα στη θητεία σας. Και τέλος, θα περιλαμβάνει η στρατηγική σας την προώθηση των ηλεκτρικών αεροπλάνων που μπορούν να δώσουν όθηση στη βιωσιμότητα των αεροπορικών μεταφορών για τις κοντινές αποστάσεις και θα μπορούσαν ίσως να δώσουν λύση στις ανάγκες των νησιών μας. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup, merci les coordinateurs. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συντονιστές ε, που έθεσαν τις ερωτήσεις. Τέσσερα λεπτά έχετε κυρία Βελάν για να απαντήσετε στο σύνολο των ερωτήσεων και να μπορέσουμε να ξανακάνουμε στη συνέχεια μια συζήτηση. Ε, φαντάζομαι όμως ότι χρειάζομαι πολύ περισσότερο χρόνο για να απαντήσω σε όλες αυτές τις ερωτήσεις γιατί θίξατε πολύ σημαντικά θέματα και θέματα νομοθεσίας, ε, θέματα ουσιώδη. Πολλοί αναφέρθηκαν στους σιδηρόδρομους. Βεβαίως και οι σιδηρόδρομοι είναι πολύ σημαντικοί για το μέλλον της Πράσινης Συμφωνίας. Έτσι λοιπόν, αφενός έχουμε την εφαρμογή του πακέτου για τους ε, σιδηρόδρομους και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε, να δούμε αν υπάρχουν διέξοδα, αν χρειαζόμαστε μέτρα για το τροχαίο υλικό, ε, για διασυνοριακή διέλευση, ε, να δούμε κατά πόσο εφαρμόζεται σωστά η δέσμοι μέτρων για τους σιδηρόδρομους. Θα το αξιολογήσουμε αυτό. Και επίσης θα εξετάσουμε και την εφαρμογή του, ε, της δέσμης μέτρων ERTMS, να δούμε και εκεί πώς ακριβώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, γιατί και αυτό θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τη συνδεσιμότητα μέσω σιδηροδρόμων. Αυτά σχετικά με τους σιδηρόδρομους. Τώρα, ίσω δεν ξέρω να αναφερθώ και λιγάκι στο θέμα του Μπρένερου. Πράγματι, την προηγούμενη εβδομάδα ε, επισκέφθηκα το διάδρομο Μπρένερο. Γιατί, διότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι των υποδομών μας στην Ευρώπη. Ε, βόρειος, ε, βορράς, νότος διάδρομος, οι Ιταλοί μεταφέρουν εμπορεύματα προς την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικός ο διάδρομος αυτός Βεβαίως ε, έγιναν πάρα πολλές συζητήσεις ε, σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω της ε, κυκλοφορίε μέσα από το διάδρομο αυτό. Δύο δι έχουν δοθεί για, το βασικό, για τη βασική σύραγγα, το Base Tunnel. Πολύ καλά πάνε εκεί οι αυστριακέ αρχές. Ε, θέλω να τις ε, συγχαρώ, γιατί είναι ε, εντός των ημερομηνιών, μέσα στο πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιες συζητήσει για τις οδούς ε, που οδηγούν, σιδηροδρομικές βασικά δυνατότητες που οδηγούν στη σύραγγα και το γερμανικό κράτος, κυρίως οι Βαβαροί, αναζητούν να βρουν τις βέλτιστες δυνατές λύσεις. Δεν είναι αρνητική, ούτε υπάρχει καθυστέρηση. Βεβαίως, ε, διαρωτώμεθα το πότε θα ξεκινήσουν οι συγκεκριμένες ενέργειες. Αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει σύραγγα και ότι αυτή δεν είναι έτοιμη. Εγώ έχω αναλάβει την υποχρέωση να το δούμε αυτό και να βρούμε την βέλτιστη δυνατή λύση πρόσβασης στη σύραγγα. Ε, Βεβαίω ε, και έχουμε μια ολόκληρη δέσμη μέτρων. Φαντάζομαι όλοι μας μιλάμε για το ίδιο. Θέλω να σας πω ότι το να επιβληθούν διόδια σε αυτή τη σύραγγα, αυτό θα ήταν η καλύτερη λύση για να ρυθμίσουμε την κυκλοφορία μέσα από τη σύραγγα. Από την άλλη όμως είπα, είναι αλήθεια ότι μονομερή μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν από τοπικές αρχές για να περιορίσουν την κυκλοφορία, αυτό δεν μπορεί να είναι αποδεκτό ε, στους ευρωπαϊκούς διαδρόμους, γιατί σήμερα είναι το Μπρένερο, αύριο θα είναι κάπου αλλού, που και αυτοί θα θεωρούν ότι περνάνε ε, από την περιοχή τους ε, πολλά φορτηγά ε, και τότε αυτό θα είναι το τέλος της εσωτερικής αγοράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα κυκλοφορίας και φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου γιατί αν ο κάθε δήμαρχος μπορεί να πει δεν μου αρέσει που περνάνε εδώ αυτοκίνητα να αναζητηθούν εναλλακτικέ λύσεις αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Εγώ αυτό είπα και σας λέω μίλησα και με τους τρεις υπουργούς και τους κάλεσα να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις έτσι ώστε να ε, ληφθούν μέτρα για την ε, εμπορευματική κυκλοφορία, κυκλοφορία φορτηγών από το Μπρένερο. Και για να είμαι ειλικρινής όμως, ε, οι αρχές του Τυρόλου ε, δεν έδειξαν ιδιαίτερη προθυμία να περιορίσουν ή να αμβλύνουν κάποιους περιορισμούς. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις συζητήσεις. Ε, ξέρετε, εγώ επειδή έρχομαι από το Κοινοβούλιο, ο συμβιβασμός μπορεί να βοηθήσει τόσο πολύ για να βελτιωθεί μια κατάσταση. Ας συνεχίσουμε λοιπόν ε, να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Ξέρω ότι δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε τη λύση. Λυπάμαι που μακρηγόρησα, αλλά ξέρω ότι αυτό ενδιαφέρει πάρα πολλούς εναλλακτικά κάψιμα για την αεροπλοεία. Αυτά εντάσσονται ε, στη δέσμη μέτρων που έχουμε κατά νου για να αφαιρέσουμε τον άνθρακα από τις αεροπορικές μεταφορές να έχουμε πιο καθαρά αεροπλάνα και όλα τα σύναφη. Πιστεύω επίσης ότι είναι ένα θέμα ε, βιομηχανικής στρατηγικής, γιατί πρέπει να συνδυάσουμε την ε, βιομηχανική στρατηγική με άλλους τομείς, έτσι ώστε να έχουμε αρκετά βιώσιμα κάψιμα για την αεροπλοεία και αυτό πραγματικά να σημαίνει κάποια διαφορά. Αυτό κοιτάζουμε και με μεγάλη μου χαρά να συνεργαστώ με τον Επίτροπο Μπρετό, έτσι ώστε να δούμε το θέμα και από πλευράς ενέργειας ενέργειας. Πώς δηλαδή μπορούμε να ενθαρρύνουμε τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων στην αεροπλοεία. Όσον αφορά κοινωνικής φύσεως θέματα, ε, το θέμα των ε, πρακτικών ε, της αυτοαπασχόλησης σε κάποιες εταιρείες. Αυτό το εξετάζουμε ε, με ενδιαφέρει. Έχω συζητήσει με κάποιους εκπροσώπους από την αεροπλοεία, όπως με την Ένωση ε, των ε, ε, Πιλότων. Βεβαίως, το πώς ακριβώς γίνεται τελικά και πώς ρυθμίζει το θέμα της απασχόλησης, αυτό είναι, θα έλεγα, και ένα εθνικό θέμα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα της ασφάλειας, να δούμε το θέμα κάτω από το πρίσμα της ασφάλειας, τις συνθήκες εργασίας, νέες συνθήκες για τους πιλότους και για τα πληρώματα. Και όταν προχωρήσουμε λιγάκι ε, θα επανέλθουμε. Αλλά όπως σας είπα, ε, βρίσκομαι σε επαφή με τις εταιρείε που προσλαμβάνουν προσωπικό ε, θέματα αυτοπασχόληση, συμβάσει και το καθεξής. Για το Brexit, ε, αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να συζητηθεί. Σε γενικές γραμμές ε, είναι πολύ σημαντικό όλα τα κρατημέλη να παραμείνουν ενωμένα στις διαπραγματεύσεις ε, για να εκπροσωπούν κοινά συμφέροντα. Εμείς βεβαίως θα εκπροσωπήσουμε τα ευρωπαϊκά ε, συμφέροντα στις διαπραγματεύσεις, συμφέροντα που θα μπορούσαν να συγκλίνουν με τα συμφέροντα του Ηνωμένου Βασιλείου όσον αφορά την οικονομική ευημερία και την ε, καλή συνεργασία ε, σε όλους τους τομείς. Όσον αφορά την αεροπλοΐα, δεν θέλω να προκαταλάβω τίποτα, αλλά θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πόσο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτή θα είναι η συζήτηση ε, και γνωρίζω ότι ο κύριος Μπαρνιέ ε, δεσμεύτηκε ε, να, έρθει, να έρχεται και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο πριν από κάθε γύρο διαπραγματεύσεων. Το ίδιο θα κάνω και εγώ. Και έχω τους συνεργάτες μου που παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις έτσι ώστε όπως σας είπα να έχουμε και να εκπροσωπούμε κοινά συμφέροντα όσον αφορά τα πολλαπλά εισιτήρια και τα δικαιώματα των ε, ε, επιβατών από τον κύριο Νταλούγκ υπάρχει αυτό το θέμα αυτή της ε, μορφή εισιτηρίων. Από την άλλη υπάρχει και το θέμα της μεταφορά δεδομένων. Αυτό πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο που να βασίζεται στην εμπιστοσύνη και πρέπει να ορίσουμε τα δεδομένα εκείνα τα οποία θα έχουν στη διάθεσή τους οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί φορείς. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το θέμα με τα εισιτήρια των πολλαπλών διαδρομών. Έχει γίνει μια σχετική μελέτη από αυτού του θέματος. Σε αυτή τη φάση έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ε, χρειαζόμαστε νομοθετικές ε, δράσεις. Αλλά πρέπει βέβαια το θέμα να το επανεξετάσουμε, γιατί όπως είπατε είναι πολύ ε, σημαντικό. Μόνο μία κουβέντα για το πακέτο κινητικότητας του κ. Λοτόφσκη η ερώτηση. Οι δέσμοι μέτρων για την κινητικότητα βεβαίως συνεπάγεται ε, βελτίωση στα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων. Αυτό είναι το σημαντικότερο και πρέπει να το στηρίξουμε. Από την άλλη, γνωρίζετε ότι ε, το Κολέγιο των Επιτρόπων, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Τίμερμανς, σε συνεργασία και σε συντονισμό με την Πράσινη Συμφωνία, καταλήξαμε στο ότι ε, όσον αφορά τις συνδυασμένες μεταφορές, την επιστροφή των φορτηγών, εκεί ενδεχομένως να μην είναι ε, τα μέτρα εναρμονισμένα με την Πράσινη Συμφωνία. Ενδεχομένως να προκύπτουν συμπληρωματικές εκπομπές και να προκύπτει και στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Αυτό είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα εμείς προβαίνουμε σε μελέτη αντικτύπου. Σε αυτή τη φάση ορίζουμε την μεθοδολογία γιατί θέλουμε η μελέτη να προσφέρει συγκεκριμένα μέτρα που θα ήταν χρήσιμα για να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις αυτού του μέτρου. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω και να σας πω και κάτι άλλο. Την Τρίτη είδα εννέα υπουργού μεταφορών από εννέα ευρωπαϊκές χώρες που ήρθαν με τις μελέτες τους και εξήγησαν σε μένα και στον κύριο Τίμερμαν τις επιπτώσεις ε, από το πακέτο κινητικότητας σε εθνικούς προπολογισμού, ε, σε ενώσεις ε, εργαζομένων και πάρα πολλά άλλα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μόλις έχουμε περισσότερα στοιχεία, ε, θα επανέλθουμε για να σας ενημερώσαμε. Ρωτήσατε σχετικά με τον χρονισμό. Ε, θέλουμε να υπάρχει καλή μελέτη αντικτύπου και αυτό σημαίνει πριν τεθούν σε εφαρμογή οι διατάξεις. Άρα δηλαδή το συζητάμε αυτό, το πόσο γρήγορα μπορούμε να προχωρήσουμε. Και τέλος το θέμα των ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένων περιοχών, η ερώτηση της κυρίας Κουντουρά ε, για τις εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Ξέρετε ότι εγώ πρέπει να είμαι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί οι άνθρωποι θέλουν τη συνδεσιμότητα για λόγους οικονομικούς, πραγματικής ζωής και γιατί όχι, και γιατί πάρα πολλοί εξ αυτών ε, ζουν από τον τουρισμό. Χρειαζόμαστε βιώσιμο τουρισμό, άρα χρειαζόμαστε συνδεσιμότητα. Προφανώς αυτό είναι αυτονόητο. Μιλήσατε και για τα ηλεκτρικά αεροπλάνα αυτό είναι το μέλλον. Αυτά τα μικρά αεροπλάνα ε, πράγματι θα συμβάλλουν ε, στο πρασίνισμα ε, και θα συμβάλλουν και στο να υπάρχει καλύτερη ψυχαγωγία και ελεύθερος χρόνος. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Επίτροπε, θα συνεχίσουμε για να σας υπενθυμίσω ότι στο θέμα της κινητικότητας, ακόμη και αν ζητούνται μελέτες, ε, ξέρετε ότι πρόκειται για μια δέσμη μέτρων που έχει μελετηθεί εδώ και τρία χρόνια και έχουμε πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να προχωρήσουμε, ακόμη και αν παράλληλα εσείς υλοποιείτε τις μελέτες σας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τέλη που δεν είναι εξαδερφός μου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ναι, είναι επίκαιρο πάντα το αστείο αυτό. Λυπάμαι κύριε Επίτροπε. αλλά θα πρέπει να αναφερθώ στα σχόλιά σας ε, για το πακέτο κινητικότητας. Αναρωτιέμαι, δεν θα ήταν πιο λογικό αν ε, Έχω ενημερωθεί σωστά. Ξέρω ότι το Συμβούλιο θα εγκρίνει σήμερα τη δεύτερη ανάγνωση. Αν έχουμε λοιπόν αυτές τις ανησυχίες και προφανώς στην νομοθεσία υπάρχουν κάποια σοβαρά προβλήματα γιατί η Ευρώπη χρειάζεται ποιοτική νομοθεσία και αν το 1 τρίτο των κρατών μελών ήδη έχουν εκφράσει αμφιβολίες Συν το ότι μάλλον θα προσφύγουμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε αν βάσει όλων αυτών των ανησυχιών και των σχολιών σας ότι υλοποιείται μελέτη αντικτύπου δεν πρέπει να δούμε αν θα πρέπει να προχωρήσουμε και όντως να ολοκληρώσουμε αυτή την νομοθετική διαδικασία και ελπίζοντα ότι αν τεθεί σε ισχύ θα παρουσιάσετε κάποια αποτελέσματα. Και τα κράτη-μέλη τελικά θα οδηγηθούν προς το να προετοιμαστούν προς αυτή τη μεταβατική περίοδο για κάτι που μπορεί όμως να αλλάξει τελικά. Αυτά, σας ευχαριστώ. Ολοκληρώστε κύριε Ντελή, ωραία. Ο κύριος Σέρτουγκ. Για ένα λεπτό έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ για όλα τα θέματα που θίξατε. Νομίζω ότι αναφερθήκατε σε όλα τα σημαντικά θέματα. Και πάλι φαίνεται ότι έχετε καλούς εμπειρογνώμονες δίπλα σας ε, από το Κοινοβουλίο. Αλλά να επαναλάβω ότι αναφέρατε σε σχέση με την υποδομή εναλλακτικών καυσίμων που είναι πολύ σημαντικό για μένα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να πετύχει τους κλιματικούς στόχους. Είναι ορθό ότι αυτή η οδηγία θα πρέπει ουσιαστικά να μεταγραφεί σε έναν μεγαλύτερο κανονισμό. Αυτή τη φήμη άκουσα αυτή την εβδομάδα. Δεύτερον, ο υψηλός αριθμός εκπομπών που έχουμε στις αστικές περιοχές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δύο στις μεγάλες πόλεις. Έχετε κάποια σχέδια σε σχέση με τις ευφυείς πόλεις, κάποια τέτοια ευφυή για τις πόλεις που θα μπορούσε να υποστηριχθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε, κύριε Σετιέν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, είπε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές σας ε, είναι ε, ανταγωνιστική κινητικότητα για το μέλλον, βιώσιμη για την αεροπλοεία Νομίζω ότι ο καλύτερο τρόπο να αποφύγουμε τι εκπομπέ εξωτερικού του άνθρακα είναι να έχουμε λιγότερη συμφόρηση και λιγότερε πτήσει. Αναφέρεται τον κανονισμό για τι χρονοθυρίδε για το θέμα αυτό, για τα σλότ. Πώ θέλετε να προχωρήσετε, από το 2012 είναι ο φάκελο αυτό. είναι πολύ παλιό. Θέλετε να τον επικαιροποιήσετε με ένα καλοπιστικό τρόπο ή θα γίνει μια αναθεώρηση εις βάθος, τι σκοπεύετε. Δεύτερον, αν σκεφτούμε τη συμφόρηση και την αεροπλοεία. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε το νεο ουρανό 2 συν. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία πιστεύετε μπορείτε να μπλοκάρετε την κατάσταση στο Συμβούλιο, γιατί εδώ και δύο χρόνια είναι μπλοκαρισμένη και δεν είναι μόνο το Γιβραλτάρο όπως γνωρίζουμε. Και πώς θέλετε να βοηθήσετε για να αναπτυχθεί η υποδομή. Γιατί αν το ένα σύστημα δεν μπορεί να συνδεθεί με το άλλο, τότε δεν θα λειτουργήσει. Πώς βλέπετε λοιπόν την ανάπτυξη. Και τρίτη ερώτηση για τα εναλλακτικά καύσιμα. Πώ θα διασφαλίσετε ότι ακόμη και αν έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή τέτοιων καυσίμων θα χρησιμοποιηθούν και στην αεροπορία, γιατί χρειαζόμαστε τέτοια εναλλακτικά καύσιμα και στην αεροπορία. Μάλιστα, κύριε Λευσόντε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε να επιμείνω εδώ στο κοινωνικό ζήτημα των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών. Πιστεύω ότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Υπάρχει το θέμα του πακέτου της κινητικότητας και των αποσπασμένων εργαζομένων στις οδικές μεταφορές και τους χαρακτηρίζει επισφάλεια. Σήμερα οι άνθρωποι αυτοί αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό. Έχουμε ακόμα πιο επισφαλείς οδηγούς που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μολδαβία, Λευκορωσία, Ρωσία, Φιλιππίνες, Καζακστάν, Σρι αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται με το χιλιόμετρο και αυτή είναι αθέμητη και πρακτική και τους οθεί να κάνουν όλο και περισσότερα χιλιόμετρα με όλου τους κινδύνους που ενέχονται. Μιλήσατε για την ασφάλεια, νομίζω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο αυτό. Δεύτερη σημαντική προβληματική, η κοινωνική κατάσταση των εργαζομένων, των πιλότων και του πληρώματος των αεροσκαφών. Όπως έχουμε ξαναπεί, έχουμε ε, κάποιες συμβάσει που υποσκάπτουν την αξιοπρέπεια και εκεί μιλάμε για απόσπαση εργαζομένων ε, για κάποιες συμβάσεις μικρής διάρκειας, ε, έμεσα καθεστώτα ε, για την πρόσληψη άνθρωποι που προέρχονται από τρίτες χώρες και μιλάμε για επισφάλεια επίσης στο πλήρωμα. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και περιμένουμε συγκεκριμένες δράσεις, κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ η κυρία Μέτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω γαλλικά. Εγώ έχω μια ερώτηση για τα μεγάλα έργα που συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε ενώ δεν έχουν πολύ μεγάλη αξία ούτε περιβαλλοντική ούτε οικονομική. Θα σας μιλήσω για το ΤΖΒ Λιόν Τωρίνο. Φαίνεται ότι η Γαλλία και η Ιταλία έχουν ζητήσει παράταση της προθεσμίας, της χρήση τη επιδότηση για να ελοποιηθεί το τούνελ ε, και έχουμε ε, μία σύμβαση για χρηματοδότηση για πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ. Ε, αυτό το θέμα ε, το συζητήσαμε, είχαμε θέσει μια γραπτή ερώτηση και η ερώτηση ήταν αν είναι ακριβείς αυτές οι πληροφορίες. Υπάρχει αυτό το αίτημα όντως για την παράταση, αν ναι, μπορείτε να μας πείτε αν ε, έχει δοθεί διθετική γνωμοδότηση για αυτή τη νέα παράταση από τον αρμόδιο φορέα, αν ε, ναι, αυτό έρχεται σε αντίθεση με την αρχή use it or lose it, έτσι δεν είναι, ε, ή ε, ουσιαστικά είναι η ουσιαστικα ειναι η διαδικασια να εξελίξει. Έχω και άλλη ερώτηση για την οδική ασφάλεια. Ξεκινήσατε τη σημερινή σας ομιλία για, σε σχέση με την επίσκεψή σας στη Στοκχόλμη. Όμως ε, δεν άκουσα να μας λέτε συγκεκριμένα μέτρα για, τον οδικό, για κάποιο οδικό χάρτη ή για διαφοροποιημένη προσέγγιση σε σχέση με τους ε, πιο αδύναμους ε, στο σύστημα, όπως ε, είναι οι ποδηλάτες, οι πεζοί. Και τελικά, ποια μέτρα θα πάρετε για το 2030. Ευχαριστώ, κυρία Τάξη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Επίτροπο Βαλεάν. Θα μιλήσω για την ευσυπλοεία. Η ευρωπαϊκή Ευσυπλοεία ε, παράγει πολλέ εκπομπέ και ρηπαίνει την ατμόσφαιρα και σίγουρα η ευσυπλοεία ρυθμίζεται από το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλία, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι στην Ένωση. Ο Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλία δεν θέτει υψηλού στόχου και συχνά μπλοκάρεται από κάποια κράτη-μέλη που δεν είναι τόσο προοδευτικά. Έχω δύο ερωτήσει, λοιπόν. ποιε συγκεκριμένε νομοθετικέ δράσει σκοπεύετε να λάβετε για να μειώσετε τι εκπομπέ στην αυσιπλοεία και υποστηρίζετε τον Επίτροπο Τίμερμαν στις προσπάθειές του για να εντάξει τον ε, τομέα της αυσιπλοείας στο σύστημα εμπορίας εκπομπών και κάτι άλλο. Ε, το τομέα ε, της ναυπηγικής μετακινείται στην Κίνα και έχουμε φτηνούς εργάτες στην Κίνα που φτιάχνουν ολόκληρα πλοία. Πιστεύω ότι οι θέσει εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να δημιουργηθούν με, την μετάβαση στις βιώσιμε μεταφορές Πώ σκοπεύετε να διατηρήσετε τις εργασίες στις βιώσιμε μεταφορές στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Σούλτς. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, χαίρομαι ιδιαίτερα που σας βλέπω στην Επιτροπή μας. Εγώ θα ήθελα να αφερθώ στους αυτοκινητόδρομους και την οδική ασφάλεια. Αναφερθήκατε σε διάφορες ιδέες και στόχους για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, αλλά συγκεκριμένη πρόταση δεν είδα. Θα μπορούσατε να μου πείτε τρει-τέσσερι συγκεκριμένε ιδέε ή προτάσει που προτίθεστε να εφαρμόσετε για την οδική ασφάλεια. Δεν χρειάζεται να επισέλθετε σε λεπτομέρειε, αλλά κάτι πιο συγκεκριμένο. Επίση, μεγάλα δήμη από τη μία και η Ήπεθρος από την άλλη. Στη νέα Ευρωπαϊκή Συμφωνία θα υπάρχουν προτάσεις σίγουρα για τα αστικά κέντρα και εκεί θα είναι διαφορετική η κινητικότητα από ό,τι στην επαρχία στις αγροτικές περιοχές. Στην Ευρώπη όμως έχουμε πολλούς δήμους ε, με λιγότερο από χίλιους κατοίκους. Και οι δήμοι αυτοί δεν έχουν τις επαρκείς υποδομές για να εφαρμόσουν τα μέτρα της Νέας Πράσινης Συμφωνίας. Επίσης, σωστά αναφέρατε την ψηφιοποίηση, αλλά και εκεί υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Και όποιος ταξιδεύει ε, οδικά από τις Βρυξέλλες για 10 λεπτά και περνάει τα σύνορα δεν μπορεί να κάνει ε, τηλέφωνα. Δεν έχουμε βασικές καν υπηρεσίες μερικές φορές, ακόμη και στις μεταφορές. Η κυρία Μπαραντίκα, σας ευχαριστώ κυρία Επιτροπέ και καλώς ήρθατε. Σας εύχομαι καλή επιτυχία και καλή τύχη και μπορείτε να υπολογίσετε στη δική μας βοήθεια και υποστήριξη. Θα ξεκινήσουμε το πακέτο της κινητικότητας που μας ε, κόστισε τεράστιες προσπάθειες, αφοσίωση, γενναιοδορία για να καταλήξουμε σε απόφαση και μας εξέπληξε αυτή η συνάντηση που είχατε. Γιατί θέλουμε να εφαρμοστεί το πακέτο κινητικότητας ακέραιο στο σύνολό του. Βέβαια, κανένας δεν συμφωνεί απόλυτα με όλα τα μέτρα. Αλλά αυτό μα ζητά ο ευρωπαϊκός κλάδος γενικώ. Και γιατί το χρειαζόμαστε, γιατί η Ολλανδία ανήγγειλε ότι από την 1η Μαρτίου θα εφαρμόσει Μονομερό κάποια μέτρα. Η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία το έκαναν ήδη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει αυτά τα θέματα προκειμένου να προχωρήσουμε στον τομέα της κινητικότητας. Τι θα κάνετε με τη μονομερή απόφαση της Ολλανδίας που από την 1η Τρίτου θα εφαρμοστεί και θα επηρεάσει το σύνολο του ευρωπαϊκού κλάδου. Κάντε παρακαλώ μια προσπάθεια να προχωρήσουμε στο πακέτο αυτό και στη συνέχεια να αναλύσουμε τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η εφαρμογή του για να το βελτιώσουμε στο μέλλον. Δεύτερον, συμφωνώ με τους στόχους που θέσαμε, αλλά πρέπει να γίνει κάποια ανάλυση που είναι κυρίως για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Γιατί ε, έχουμε αύξηση στις διασυνοριακές περιοχές ε, των ε, εκπομπών Πώς θα απαιτήσετε από τα κράτη-μέλη να τηρήσουν επιτέλους την εκτέλεση ε, και τις προθεσμίες των ε, σχεδίων TNT, των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Πώς αλλιώς θα υλοποιήσουμε τους στόχους. Επίσης, την αλλαγή του θερινού ωραρίου. Ήδη έχουμε εγκρίνει την οδηγία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Συμβούλιο ε, θα λάβει κάποια θέση, θα προχωρήσει επιτέλους το θέμα της αλλαγής της ώρας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κρίμα που μερικές φορές δεν έχουμε αρκετό χρόνο για να ολοκληρώνουμε τις παρεμβάσεις μας. Και γι' αυτό κάποιοι συνάδελφοι δεν, μπόρεσαν, δεν πρόλαβαν να δώσουν όλες τις πληροφορίες. Για τον Μπρένερο, για παράδειγμα, κάποιοι επιχειρηματίες εξαιρούνται από τους περιορισμούς και η Ιταλή Παραγωγή λένε μην ανησυχείτε, εμείς μπορούμε να αναλάβουμε αυτό το έργο που κάνουν οι τέλη μεταφορείς για σας. Οπότε το θέμα είναι όλοι αντιλαμβανόμαστε τους λόγους των υπόλοιπων, γνωρίζουμε τους λόγους που έχουν οι Τυρολέζοι και γνωρίζουμε και τα επιχειρήματα της ιταλικής πλευράς για τον Μπρένερο. Ξέρουμε ότι οι Ιταλοί δεν σέβονται το χρονοδιάγραμμα και τις προθεσμίες και προσπαθούμε, ε, προσπαθήσαμε προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε και ένα χρόνο νωρίτερα ε, τα έργα για τον Μπρένερο, αλλά οι τελικές κυβερνήσεις, η, η τωρινή, η επόμενη, δεν ξέρω αν είναι έτοιμες να το στηρίξουν, αλλά είναι και θέμα χρόνου, γιατί όλοι οι διάδρομοι των διευρωπαϊκών δίκτυων μεταφορών θα επηρεαστούν από αυτήν την απόφαση και ελπίζω να βρούμε λύση, θέλουμε να βρούμε λύση μέχρι το 2028, ίσως και το 2027. Μακάρι. Αλλά είναι παράδοξο να έχουμε υποτίθεται ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και προσώπων και να προσκρούμε σε τέτοια εμπόδια. Κυρία Νάτεγκαλ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, καλώς ήρθατε. Εγώ θα μιλήσω για τις Διεθνείς συμφωνίε για τις ενέργειε Μεταφορές. Το 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε εντολή να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια συνολική συμφωνία για την αεροπορία με το ΟΜΑΝ. Έχουν ήδη λάβει χώρα δύο γύρι διαπραγματεύσεων. Βέβαια, η βιωσιμότητα είναι και δική σας προτεραιότητα, όπως φαίνεται. Και ελπίζω να το τονίσατε. Η Ευρωπαϊκή Αεροπλοεία επίσης θέλει να συμβάλλει ε, δικαίως στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Και τώρα, δεδομένου το ότι η αεροπορία είναι ένας παγκόσμιος κλάδος, δεν είναι μόνο ευρωπαϊκός και χρειαζόμαστε θεμητό ανταγωνισμό και από τρίτες χώρες. Ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ όρων των αεροπορικών εταιριών, αυτό είναι απαραίτητο ε, απαραίτητη προϋπόθεση. Σκέφτεστε λοιπόν να συμπεριλάβετε και μια περιβαλλοντική ρήτρα με συγκρίσιμες προδιαγραφές όπως παρουσιάζεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στις, ε, εταιρείες, στις συμφωνίες ενέργειων μεταφορών που θα έχουμε τώρα με το ΟΜΑΝΙ και στις μελλοντικέ ε, συμφωνίες για την αεροπορία που θα συνάψετε με τρίτες χώρες. Σας ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ δυστυχώς θα πρέπει να φύγω. Θα με αντικαταστήσει ο αγαπητός συνάδελφος κύριος Σούλτς. Πάντως, ε, πριν φύγω θα ήθελα να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξαναθέσει το πακέτο για τις εμπορευματικές σιδηροδρομικές μεταφορές. Επίσης, τι θα γίνει με την Ευρωβινιέτα, θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις, ε, ναι και πότε, αν ναι. Επίσης, ε, μιλήσαμε πολύ για την αεροπορία. Θα έχουμε τον κοινό ευρωπαϊκό ουρανό, αλλά είναι και πρόβλημα η χρηματοδότησή του. Μιλούμε για το φόρο της κυροζήνης. Εννέα χώρες προωθούν αυτό το φόρο θα αισθενιστείτε αυτή την πρόταση. Σε ό,τι αφορά το πακέτο της κινητικότητας, το Κοινοβούλιο έκανε το καθήκον του και θα συνεχίσουμε, θα περάσουμε στη δεύτερη ανάγνωση. Και έχετε δίκιο που ε, αναφέρεστε στις αξιολογήσεις, αλλά το κοινοβουλευτικό έργο θα πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ φεύγω, αλλά θα σας αφήσω στα επιδέξια χέρια του κύριου Σούλτς. I'm waiting for guidance from Mr. Schulz. Περιμένω ε, κάποιες οδηγίες από τον κύριο Σούλτς. So, wir machen, weil wir schon ein bisschen äh, vorangeschritten Λοιπόν, έχει ε, προχωρήσει η ώρα, ε, γι' αυτό να προχωρήσουμε λίγο γρήγορα. Η κυρία Πάουλους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και την Επίτροπο. Λυπάμαι, αλλά θα επανέλθω στο ζήτημα του Μπρένερου, γιατί πραγματικά δεν το καταλαβαίνω. Είπατε ότι προτείνετε να αυξήσετε τα διόδια ως λύση και είπατε ότι ταυτόχρονα δεν θα δεχτείτε μονομερή περιφερειακά μέτρα. Κατά τη γνώμη μου, η αύξηση των διοδίων είναι μονομερές περιφερειακό μέτρο. Οπότε πώς, εσείς πώς το, θα, αλλιώς θα το περιγράφατε δηλαδή. Δεν ήμουν παρούσα δυστυχώς στο Τυρόλο όταν πήγατε στη συνάντηση και δεν βρήκα τίποτα στην ενημέρωση. Ποια είναι τα μέτρα που προτείνατε και που έχετε αναφέρει επανειλημμένως. Τα αναφέρετε όμως γενικά, αλλά χωρίς λεπτομέρειες. Με ενδιαφέρουν όμως συγκεκριμένα ποια μέτρα έχετε κατά νου. Επίσης, για τα εναλλακτικά καύσιμα, πιστεύω ότι αν υπάρχει ένας τομέας που μπορούμε να έχουμε βιώσιμα εναλλακτικά καύσιμα στην Ευρώπη και γενικώ, ο τομέας αυτός είναι περιορισμένος, γιατί έχουμε και την ανάγκη επισητισμού και την ανάγκη κάποιων ε, ζωνών ε, φύσης, ε, φυσικών χώρων. Οπότε ίσως θα έπρεπε να περιορίσουμε τα εναλλακτικά καύσιμα μόνο σε μερικές περιπτώσεις στην αεροπορία. Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ε, να τηρείτε το χρόνο. Ε, ευχαριστώ για την Επίτροπο, γιατί θα μείνει λίγο παραπάνω, το δέχτηκε. Παρ' όλα αυτά, να τηρείτε το χρόνο, σας παρακαλώ. Κυρία Γκαρσία Μουνιός. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ και την Επίτροπο. Επανέρχομαι στο θέμα των δικαιωμάτων και των κοινωνικών προτύπων των εργαζομένων στην αεροπορία. Ένα θέμα που συνάδει και με την ανάγκη της ασφάλειας των αερομεταφορών που είπατε. Είναι ένα θέμα διασυνοριακό σίγουρο. Δεν είναι εθνικό ζήτημα. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν πανευρωπαϊκές λύσεις συνολικέ με συγκεκριμένε δράσει, γιατί οι εργασιακέ συνθήκε μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια, την εναέρεια και την ασφάλεια των επιβατών. Σίγουρα συνεργάζεστε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Ενέργειας Κυκλοφορίας. Συζητάτε όμως για τα νέα συμβόλαια που έχουν γίνει πολύ της μόδας σε κάποιες αεροπορικές εταιρείες, κυρίως στις low cost εταιρείες, γιατί πρόκειται για επισφαλείς θέσεις εργασίας, για ψευδοαπασχολούμενους, για συμβάσεις μηδενικών ορών. Μερικές φορές το πλήρωμα αναγκάζεται ακόμη και άρρωστο να εργαστεί από φόβο μην απολυθεί ή να μην ξαναδουλέψει λαμβάνετε υπόψη όλους αυτούς τους κινδύνους που δεν είναι μόνο κοινωνικο-οικονομικοί αλλά και θέμα ε, εναέρειας ασφάλειας. Ε, αυτά τα συμβόλαια δημιουργούν πολλούς κινδύνους. Επίσης, πώς θα αποφύγουμε τη στρέβλωση ανταγωνισμού από κάποιες αεροπορικές εταιρείε με το κοινωνικό dumping που επιβάλλουν και χρησιμοποιώντας κάποια νομικά κενά της ενωσιακής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νόβακοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις. Ξέρω ότι σχολιάσατε επανειλημμένο στο πακέτο κινητικότητας, αλλά έχω και εγώ μια ερώτηση που μέχρι στιγμής δεν έχει καλυφθεί. Είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει στοχευμένη νομοθεσία ε, όπως ε, η επιστροφή των φορτικών άδειων γιατί φαίνεται ότι μιλούμε με πάθος για τις οικολογικές, φιλοπεριβαλλοντικές ιδέες και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, αλλά πώ συνάδει ε, με τη Νέα Πράσινη Συμφωνία αυτή η επιστροφή των άδειων φορτηγών. Δεύτερον, η πρόταση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο του κυρίου Μισελ λέει ότι ε, γίνεται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όμως διαπιστώνουμε 35% περικοπές στο συνδέοντα στην Ευρώπη σε σχέση με την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που τους ή άλλως είναι 10% λιγότερο από την παρούσα πρόταση. Θα αντιδράσετε σε αυτή τη δραστική περικοπή του μηχανισμού συνδέοντα στην Ευρώπη που πόρο απέχει και από τις φιλοδοξίες μας για την ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φέρμπερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτά τα ξεκάθαρα λόγια που είπατε στο Τυρόλο. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ε, μία Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβάλλει κυρίως το ευρωπαϊκό στοιχείο. Αυτά που είπε στον Άλφος από την Ιταλία είναι σωστά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν ε, κάτω από την πρόφαση ή την δικαιολογία του περιβάλλοντος, οι Τυρολέζοι ε, κάνουν διαφήμιση στην Ιταλία και τη Γερμανία ότι αυτοί μπορούν να βρουν τη λύση γιατί αυτοί δεν θίγονται από τα μονόπλευρα μέτρα. Οι Βαβαροί και οι Ιταλοί δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Βέβαια, τι σχέση έχει αυτό με το περιβάλλον, κανείς δεν μπόρεσε να μου το εξηγήσει και γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ερωτήσω πότε ακριβώς ε, προτίθεστε να άρετε αυτά τα μονομερή μέτρα ε, και προτίθεστε να καταγγείλετε και την πόλη του Τυρόλου για όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φέρμπα. Ε, κύριος Βιτάνοφ. Οι προσπάθειες της κυρίας Βαλεάν και όλες της Κομισιόν για μια βιώσιμη κινητικότητα είναι αξιέπαινες, όμως θα πρέπει να κάνουμε μεγάλες προσπάθειες και να δώσουμε μία συνέχεια. Λέμε ότι θέλουμε ένα πέρασμα προς καθαρές μεταφορές και ταυτόχρονα δεχόμαστε ότι τα βαρέα οχήματα να γυρνάνε άδεια κάθε 8 εβδομάδες. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μία αξιολόγηση της ε, κατάστασης ε, πριν να λάβουμε αποφάσεις. Και επίσης ε, θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση που συμπληρώνει την ερώτηση του κυρίου Ντάνιελσον, η Ευρωπαϊκή Αεροπορία. Διαπιστώνουμε τα τελευταία χρόνια ότι έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό στην αεροπορία και κάποιες ε, χειρότερες συνθήκες εργασίας ε, και λιγότερη ασφάλεια. Νομίζω ότι η Κομισιόν ε, θα πρέπει να προτείνει νέα νομοθεσία για να θέσει τέλος στις ψευδοσυμβάσεις των ανθρώπων που πληρώνουν ίδια τις εισφορές τους. Βλέπω μετά το Brexit, λέει ο Πρόεδρος, έχουμε και νέους συναδέλφους. Μία εξ αυτών η συνάδελφος Κλάμπ. Παρακαλώ πολύ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Στα ρουμανικά θα μιλήσω. Σας ευχαριστώ. Είναι πολύ φιλόδοξο ο τομέα των μεταφορών. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε μια πολύ σημαντική πτυχή και συγκεκριμένα στις ανάγκες να λάβουμε περισσότερα μέτρα προκειμένου να πετύχουμε τον στόχο της καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής, ε, να έχουμε βιώσιμη μετάβαση και να αντιμετωπίσουμε και εδω κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα. Ξέρετε ότι έχουμε πολλές περιοχές στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και πολλοί πολίτες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στερούνται του δικαιώματος στην κινητικότητα. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε την εδαφική συνοχή αλλά και την κοινωνική ένταξη και μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στο εσωτερικό των περιοχών αυτών. Θα συνεργαστείτε με τα κράτη-μέλη, θα τα υποστηρίξετε. Σήμερα έχουμε και τη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συζητηθεί ο μελλοντικό προπολογισμό. Και εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ποια θα είναι η δική σα θέση απέναντι στο μέσο συνδέοντα την Ευρώπη ω κύριο μηχανισμό χρηματοδότηση καθώς ε, ισχύει το γεγονός ότι χρειάζονται επενδύσει στην ε, μελλοντική περίοδο. Σα ευχαριστώ. <clears throat> Και για σας όμως παρακαλώ η τήρηση του χρόνο αγόρευσης. Η επόμενη συνάδελφος, συνάδελφος Ναχτιγκάλ. Όχι, λάθος τον κατάλογο. Η κυρία Βίρκουνεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστούμε για αυτά που μας είπατε. Ε, νομίζω ότι η αφαίρεση του άνθρακα από τις μεταφορές είναι η μεγαλύτερη πρόκληση κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας και όπως ξέρετε είναι καθοριστικό στοιχείο της Πράσινης Συμφωνίας. Παράλληλα καλούμεθα να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Αναφέρατε ορισμένες πολύ ενδιαφέρουσες πρωτοβουλίες. Είπατε ότι τώρα προετοιμάζεται κατά κάποιον τρόπο το πρασίνισμα των εμπορευματικών μεταφορών. Ε, μένα θα με ενδιαφέρε να ακούσω κάτι παραπάνω, δηλαδή ε, ποια είναι τα βασικά στοιχεία αυτού του πρασινίσματος, ε, τι μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτό το πρόγραμμα ε, και κατόπιν αναφερθήκατε και σε σιδηρόδρομους, σε διαδρόμους σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών και νομίζω ότι με αυτά τα νέα προγράμματα θα υπάρχουν επιπτώσεις και στα προγράμματα στα διευρωπαϊκά προγράμματα. Ευχαριστούμε την κυρία Φερκούνεν, ο κύριος Φερναντίνιο. κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο να γίνονται αυτέ οι συζητήσει με εσά. Ε, Κυρίω θα ευχόμουν αυτό να γίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Έχω πάρα πολλέ ερωτήσει ε, να κάνω, αλλά θα προσπαθήσω να τηρήσω το χρόνο μου και θα κάνω μία μόνο ερώτηση. Αυτό που με απασχολεί πάρα πολύ, το θέμα τη Ευρωβινιέτα. Ε, στην Ευρώπη πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα από του σημαντικότερου στόχου και το πρασίνισμα, η προστασία του περιβάλλοντο ο αγώνα κατά τη κλιματική αλλαγή. Υπάρχει όμως μια διάταξη πάρα πολύ σημαντική που θα μπορούσε να βοηθήσει πολύ το περιβάλλον, δηλαδή να μειωθούν οι εκπομπές, να βελτιωθεί η οδιακή ασφάλεια, ε, να έχουμε εναλλακτικέ ε, μεταφορές, ε, παραδείγματο χάρη σιδηροδρομικές μεταφορές και όλα αυτά έχουν μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο και κανείς δεν ξέρει πια πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν τι ακριβώς προτίθεται να κάνει. Εσείς προτίθεστε να έρθετε σε αντιπαράθεση με τις χώρες εκείνες οι οποίες ε, μπλοκάρουν αυτή την τόσο σημαντική πρόβλεψη. Ε, τι ε, πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει έτσι ώστε να υπάρξουν διάλογοι και να δημιουργηθούν και κάποιες σχέσεις έτσι ώστε εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή να έχουμε μια τόσο σημαντική ρύθμιση για την Ευρωβινιέτα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φουρόρε παρακαλώ επόμενος συνάδελφος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω σε ένα θέμα το οποίο ήδη το έχουμε θίξει. Ε, πρόκειται για τις ε, μειονεκτούσες ε, περιοχές που αυτή τη στιγμή υφίστανται διπλή τιμωρία έξω από, τις, από τους μεγάλους διαδρόμους και δεν έχουν και κονδύλια για την απαραίτητη υποδομή. Δηλαδή προτιμάει κανείς να κάνει επενδύσεις στους δρόμους και όχι στους συνδρόδρομους. Σύμφωνα με τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Επιτροπής μέχρι το 2050 οι περισσότερες μεταφορές ε, μικρής μεσαίας απόστασης πρέπει να γίνονται με σιδηρόδρομους. Στην Ιταλία έχουμε κατά νου την Καλαβρία, την Σικελία, την Βασιλικάτα, αλλά ήδη τώρα ε, δεν υπάρχει διασύνδεση με το Βορρά και με την Ευρώπη ε, παρά μόνο χρησιμοποιώντας το αεροπλάνο. Θέλω λοιπόν εσείς τι προβλέπετε για να κινητροδοτήσετε την χρήση των σιδηροδρόμων για αποστάσεις μικρές και μεσές. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος ε, και τελευταία συνάδελφος Βόλο. Καλημέρα σας, ε, κύριε Επίτροπε. Ε, εγώ ζήσετε το λόγο γιατί θέλω να σας επισημάνω τις ε, περιφερειακές ε, περιοχές της Ευρώπης. Κατά τους επόμενους μήνες επιτέλους θα είναι δυνατόν να ε, εξετάσουμε κάποια θέματα των διευρωπαϊκών δικτύων. Στην Ευρώπη, στην Ιταλία και σε άλλες περιοχές υπάρχουν κάποιες περιοχές που έχουν μεγάλα προβλήματα και δεν έχουν αυτοκινητόδρομους, δεν έχουν σιδηρόδρομους και η μόνη λύση για να συνδεθούν είναι το αεροπλάνο. Πολλοί επισκέπτονται την Ιταλία το καλοκαίρι και θέλω να σας ρωτήσω, στην Νότια Ιταλία πώς θα έρθετε στο Ποζιτάνο, στη Νάπολη, στη Πούλια, ε, σε πολλές περιοχές. Ε, πώς θα το κάνετε αυτό με το αυτοκίνητό σας, ε, φαντάζομαι έτσι προτίθεται να το κάνετε, αλλά τις ίδιες ακριβώς διακοπές θα μπορούσε κανείς να κάνει και με δημόσιες μεταφορές. Όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα, Αγαπητοί Επίτροπε, μήπως ε, μπορούμε να υπολογίζουμε στη δική σας τη βοήθεια, έτσι ώστε να γίνεται σαφής αναφορά στις υποδομές ε, των απομακρυσμένων περιοχών. Και ίσως θα μπορούσα να σας ε, συναντήσω στην Ιταλία να κάνουμε μαζί μια περιήγηση σε όλες αυτές τις περιοχές που σας ανέφερα. Αν το κάνουμε αυτό με ένα δημόσιο μέσο μεταφοράς, ε, τότε μόνοι σας θα έχετε την ευκαιρία να κρίνετε αν αυτά που λέω είναι σωστά ή όχι. Ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Ε, κύριε Επίτροπε, έχετε πολλές ερωτήσεις. Ε, εν μέρη αυτές ε, είναι και πολύ εξειδικευμένες, είναι και σαφείς. Δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να απαντήσετε σε όλες. Παρακαλώ όμως, ε, έχετε το λόγο. Ε, μισό λεπτό όμως, είδα ότι άλλη μία συνάδελφος ζήτησε το λόγο, κυρία Ντεπανή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία ε, και εγώ να κάνω μία ερώτηση. Ε, κοιτάξτε, κύριε Επίτροπε, θέλω να θίξω ένα θέμα στο οποίο ε, δεν εμβαθύνατε. Σχετικά με την κινητικότητα, με τους, στους αυτοκινητόδρομους, ξέρουμε ότι τα εκπομπές ε, σε μεγάλο βαθμό από αυτό το, αυτή την κινητικότητα επιβαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν βέβαια ε, πάρα πολύ καλά παραδείγματα. Ε, η δική σας στρατηγική ποια ακριβώς είναι έτσι ώστε να ασκηθεί λίγο μεγαλύτερη πίεση στις πόλεις και στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αστική κινητικότητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την τελευταία ερώτηση. Κύριε Επίτροπε, τώρα έχετε το λόγο. Well, Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. ουσιαστικά φύγουν πάρα πολλά θέματα και πολύ σημαντικά θέματα για το μέλλον της πολιτικής μεταφορών. Πολύ επανήλθατε στο θέμα του πακέτου κινητικότητας. Ξέρετε ότι συνεχίζονται οι διαδικασίες και δεν μπορούμε να σταματήσουμε την νομοθετική διαδικασία. Επομένω έτσι έχουν τα πράγματα. Αναλόγως ε, με το τι θα προκύψει από τη μελέτη αντικτύπου, ε, θα δούμε αν ε, θα έχουμε στοχευμένη νομοθεσία για να αντιμετωπίσουμε να διορθώσουμε κάποια ζητήματα. Πολλοί μίλησαν για την οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων χρειαζόμαστε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο ε, σημεία μέχρι το 2025 ε, για την ε, φόρτιση και θα πρέπει να δούμε τι ρυθμιστικά μέτρα θα απαιτούνται περαιτέρω προκειμένου να αναλύσουμε τον αντίκτυπο των ε, κανονιστικών στόχων σε ό,τι αφορά τα σημεία της φόρτισης. Θα πρέπει να δούμε τι θα σημαίνει αυτό και για τους φορολογούμενους. Επίσης, ε, θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να αναπτυχθεί ε, σε σχέση με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εντό του σημερινού ηλεκτρικού συστήματο. Τώρα, αστική κινητικότητα. Είχαμε κάποια τελευταία ερώτηση σχετική οι υπηρεσίε άρχισαν την αξιολόγηση για το πακέτο της αστικής κινητικότητας από το 2013 για να εξετάσουν αν είναι κατάλληλο ε, το πλαίσιο για να εξυπηρετήσει το σκοπό. Μέχρι το Μάιο θα έχετε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής, έτσι λοιπόν ε, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση. Προκαταρκτικά, ποιο είναι το πόρισμα. Ότι δεν έχουμε τα αποτελέσματα που αναμέναμε από το πλαίσιο, γιατί έχουμε μια κατάσταση που είναι πολύ διαφοροποιημένη σε τοπικό επίπεδο και εξαρτάται από τη βούληση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Και επίσης οι πόλεις που ε, ανήκουν σε αυτό το πλαίσιο εξαρτώνται πολύ από τους δείκτες που έχουμε για την αστική κινητικότητα. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βάλουμε νέα βασικά στοιχεία στην νέα ευφυή e στρατηγική για τις ε, μεταφορές. Ε, έτσι λοιπόν θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Έχουμε πολλά να πούμε και αν το επιθυμείτε μπορούμε να αφιερώσουμε μια ειδική συζήτηση για την αστική κινητικότητα γιατί δεν ε, προλαβαίνω να καλύψω τώρα όλα τα σημαντικά πράγματα. Τώρα για την ε, Λιόν Τωρίνο προετοιμάζουμε μια απάντηση στην επιστολή σας η απάντηση θα επιβεβαιώσει ότι η σημερινή συμφωνία για τις επιδοτήσεις ίσχυε μέχρι την 31 Δεκεμβρίου πέρσι. Ε, όμως, ε, καθώς έχουμε πολλούς μήνες καθυστέρηση, οι δικαιούχοι ζήτησαν παράταση της συμφωνίας και οι υπηρεσίε μου κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εν λόγω έργο σέβεται τις προϋποθέσεις για την παράταση και τώρα διαπραγματευόμαστε με τους δικαιούχους του έργου για την ακριβή διάρκεια και την πιθανή παράταση για το παιδί εφαρμογή και την εφαρμοστέα δράση. Αλλά θα λάβετε και την απάντηση σύντομα. Για το θέμα της ασφάλειας, κύριε Λεσαντέ, αναφέρατε και πάλι το θέμα της δικαιοσύνης και του ανταγωνισμού από τρίτες χώρες. Εδώ είστε? Όχι. Ήθελα να πω ότι έχουν αυξηθεί ε, οι αριθμοί των αδειών για τους Ρώσους ε, οδηγούς ε, φέτος στη Γαλλία και αυτό μας δείχνει ότι υπάρχει αυξημένη ανάγκη και ότι οι εθνικές αρχές θα πρέπει να σκεφτούν πως αυτές οι άδειες που είναι εθνική αρμοδιότητα προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού για τους Ευρωπαίους οδηγούς. Για την πρόταση για τις χρονοθυρίδες, νομίζω ότι είπα ήδη ότι θα το εξετάσουμε. Τώρα το πρασίνισμα των θελάσσιων μεταφορών. Σήμερα το απόγευμα ξεκινά η εβδομάδα για την ευσυπλοεία και ήδη θα συζητήσουμε τους αρμόδιους σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και με τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας γιατί πρόκειται για έναν παγκόσμιο κλάδο και θα πρέπει να πρασινίσουμε τα πλοία και τους λιμένες μας για να είμαστε ανταγωνιστικοί. Νομίζω ότι συζητάμε ήδη κάποιες από τις ιδέες που είναι επιτάπτους αλλά φυσικά θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και η στρατηγική θα αντικατοπτρίζει ένα όραμα για τον θαλάσσιο τομέα για τον ναυτιλία. Τώρα, ε, για το ΕΤΕΣ ε, θα πρέπει το σύστημα εμπορίας εκπομπών επίσης να συντονιστεί ε, στα πλαίσια του ΔΟΝ. Και μιλάμε για ένα καλάθι μέτρων και εδώ έχουμε τον Μπρένερ. Θέλουμε τα μέτρα στο καλάθι Όπως ε, σας είπα, έχουμε τον τρέχοντα κανονισμό για να μειώσουμε ε, το σύστημα που προκαλεί συμφόρηση. Και είπε και η κυρία Παραντικά, ε, αναφέρθηκε στα σύνορα. Και αυτό είναι ένα θέμα που υπάρχει στη μέτρων κινητικότητας και μας ανησυχεί. Γιατί όταν έχουμε ένα φορτηγό που επιστρέφει για χώρες μη Σέγγεν σημαίνει ότι θα έχουμε ουρές και συμφόρηση στα σύνορα. Έτσι λοιπόν δεν ε, μιλάμε μόνο για το θέμα της ανάπτυξης των υποδομών, αλλά είναι και θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τη συμφόρηση και την κυκλοφορία. Για να επανέλθω στον Μπρένερ. Μιλήσαμε για τα διόδια Κάποια από τα μέτρα εδώ τα συζητήσαμε. Είχαμε εναλλακτικέ προτάσεις, είχαμε το σύστημα μεταστορών και την ψηφιοποίηση των διαδρόμων για να μειώσουμε τη συμφόρηση, να ε, έχουμε εναλλακτικέ για τι οδικέ μεταφορέ, να συνδυάσουμε οδικέ και σιδηροδρομικέ μεταφορέ. Έχουμε συντονισμένη ανάπτυξη υποδομών για εναλλακτικά καύσιμα, προκειμένου να προωθήσουμε την καθαρή κινητικότητα στο διάδρομο και διαλέγω εδώ κάποια γιατί φυσικά λεπτομερώς αυτά θα τα συζητήσουμε με τα τρία μέρη για να καταλήξουμε στο ότι είναι αποδεκτό σε όλους και να έχουμε ταχύ εφαρμογή. Φυσικά ε, να έχουμε και το Ευρωπαϊκό ε, Σύστημα Διαχείρισης Συνδροδρομικών ε, Μεταφορών, επίσης να έχουμε φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τον δίζελ και να μειώσουμε τα κίνητρα για την αγορά αυτοκινήτων δίζελ, ελέγχου στα σύνορα, να μην έχουμε ελέγχους στα σύνορα, να έχουμε διαλειτουργικότητα στους σιδηροδρόμους Πολλά μέτρα έχουμε επί χάρτου και είναι γνωστά αυτά στα μέρη ε, και αφού θα ξεκινήσουμε εκ νέου τη συζήτηση είμαι βέβαια ότι θα επανέλθουμε σε εσά με περισσότερες λεπτομέρειες και συμφωνίες. Αλλά όπως ε, σας είπα, τα διόδια για όλο το διάδρομο, για το διάδρομο Μπρένερ, ε, είπα ένα διόδιο που θα φορά το διάδρομο Μπρένερ. Δεν μίλησα μόνο για την αυστριακή πλευρά. Θα πρέπει να έχουμε μια καθολική λύση για το διάδρομο. Όχι κατακαιρματισμένη λύση ανάλογα με τις χώρες. Και υπήρχε μια ερώτηση από τον κύριο Φέρμπερ. Ναι, σκοπεύουμε να πάρουμε μέτρα. Και σε αυτό το στάδιο κάνουμε ανάλυση για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για την οδική ασφάλεια. Πρέπει να δούμε πώς ο Γενικός Κανονισμός για την ασφάλεια, για τα οχήματα και τις υποδομές εφαρμόζεται. Να δούμε εδώ ποια είναι η προσθεμένη αξία που θα φέρει. Και φυσικά σχεδιάζουμε μια αναθεώρηση συμπληρωματική με την οδηγία για την άδεια οδήγηση Φέτος. Και πάλι έχουμε ένα καλάθι μέτρων για να βελτιώσουμε την οδική ασφάλεια. Θα σας διαβεβαιώ ότι έχουμε συγκεκριμένα πράγματα κατά νου δεν θέτουμε απλώ ένα στόχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πολλοί αναφέρθηκαν στην Ευρωβινιέτα και στον Ευρωνέο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Νομίζω ότι όλοι οι υπουργοί, τουλάχιστον μία φορά από τότε που ανέλαβα ως επίτροπος, έχουν συναντηθεί μαζί μου και σε κάθε συνάντηση αυτά τα δύο θέματα συζητήσαμε. Κάθε φορά τα ανέφερα γιατί εξαρτώνται από τους υπουργού και νομίζω ότι είμαι σε καλό δρόμο. Έχω την πεποίθηση ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στον Ευρωπαϊκό Ουρανό Ιδίω επειδή έχουμε αυτή την ε, έκθεση της Επιτροπής των Σοφών για το Συμβούλιο, για το πώς να προχωρήσουμε και στο τελευταίο Συμβούλιο από τη Φιλανδική Προεδρία παραδέχτηκε το γεγονός και δεσμεύτηκε να συνεχίσει το έργο για τον Ευρωπαϊκό Ουρανό. Αυτό είναι το ένα. Τώρα για την Ευρωβινιέτα, τι κάνω. Δημερός προσπαθώ να εντοπίσω που είναι τα σημεία εμπλοκής για τις διάφορες χώρες. Όμως, ε, εγώ είμαι δεσμευμένη στην αρχή και νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωβινιέτα. Αλλά ας δούμε την αποδεκτό στο στάδιο αυτό και αν μπορούμε να απεμπλοκάρουμε την κατάσταση. Ελπίζω ότι θα ξανανοίξει τουλάχιστον η συζήτηση κατά την κρατική προεδρία. Και ελπίζω ότι η Γερμανική Προεδρία θα μας παρουσιάσει ένα είδος ευρωβιγγέτας ε, που θα είναι αποτελεσματική για όλα τα κράτη-μέλη, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές πρακτικές, τις ευαισθησίες, τις παραδόσεις κτλ. Επομένω και η Ευρωβινιέτα και ο Νέο Ευρωπαϊκό Ουρανό είναι υψηλά στο θεματολογιό μα. Ε, τώρα, σήμερα αρχίζει η συζήτηση και για τον προπολογισμό. Γνωρίζουμε βέβαια ότι πέρα από τις ε, φιλοδοξίες που είχαν η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο, τώρα το ίδιο πραγματευτικό κουτί προτείνει για το ΣΕΦ ο μηχανισμό συνδέεται στην Ευρώπη. 21,4 δισεκατομμύρια, δεν είμαι σίγουρη, αλλά μόνο 1,5 για την κινητικότητα. Γιατί ε, νομίζω ότι είναι απώλεια αυτό. Έχουν επενδυθεί πολλά στις υποδομές. Όμως από την άλλη, θέλω να μοιραστώ μαζί σας την ιδέα ότι οι διαπραγματεύσει θα πρέπει να ολοκληρωθούν κάποια στιγμή εν ώψη του πρώτου ΣΕΦ 2 την ε, σχετική υποβολή προτάσεων που είναι στο πρώτο εξάμεινο του 2021. Πρέπει λοιπόν ε, ταχύτατα να διαπραγματευτούμε πριν από αυτή την ημερομηνία, γιατί η μεγαλύτερη καθεστάριση θα είχε αποτέλεσμα αναβολή των επενδύσεων στις μεταφορές. Κυρία Πλούμπ, αναφέρατε στο, στο θέμα της συνοχής στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι σημαντική σχέση με το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο για να διατηρήσουμε όλα τα χρηματοοικονομικά εργαλεία τα οποία προβαίνουν σε ανάμιξη, σε blending. Ε, γιατί έχουμε κάποιες ε, περιοχές και χώρες ε, που ε, είναι σε χαμηλότερη ανάπτυξη και κυρίως στην Ανατολική Ευρώπη. Είναι σημαντικό λοιπόν να χρησιμοποιούνται τα χρήματα του ΣΕΦ ε, για τις υποδομές, αλλά χρειαζόμαστε και χρήματα από τα περιφερειακά ταμεία για τη συνοχή. Έτσι λοιπόν είμαι σίγουρη ότι οι χώρες ε, αυτές θα ασκήσουν πίεση για να έχουμε ένα τέτοιο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εγώ νομίζω είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί και το δίκτυο διευρωπαϊκό, το διευρωπαϊκό δίκτυο για τις μεταφορές και για τις χώρες που καθυστερούν. Και πώς θα βοηθήσουμε, θα βοηθήσουμε ε, με την εργή του κυρίου Ρικέ, με το streamlining, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θέλω και πάλι όμως να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να ανοίξετε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, γιατί πιστεύω ότι το streamlining είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να βοηθήσει τα έργα υποδομών που έχουν τεράστιες καθυστερήσεις αυτή τη στιγμή. Ίσως να υπήρξαν και άλλες ερωτήσεις. Τις έχει καταγράψει η ομάδα μου και αν είναι κάτι που παρέλειψα, θα επανέλθουμε λεπτομερέστερα σε εσά και παρακαλώ, μπορείτε και να μου γράψετε, να στείλετε ερωτήσεις στην Κομισιόν και θα σας απαντήσουμε λεπτομερέστερα για τα θέματα που σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Και δεσμεύομαι εδώ κύριε Πρόεδρε να έρθω όποτε με προσκαλέσετε, για να έχουμε ένα μόνιμο διάλογο μεταξύ Κομισιών και Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε ε, και εξ των συναδέλφων. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ ε, που συζητήσαμε για διάφορα θέματα και εσείς η ίδια για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα βρισκόσασταν στη δική μας τη θέση. Νομίζω λοιπόν ότι για σας είναι απόλυτα κατανοητό ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα μια ουσιαστική και συχνή ανταλλαγή απόψεων όπως συνέβη και κατά το παρελθόν. Σας ευχαριστώ πολύ. So, Παρακαλώ όσους ε, είναι όρθιοι, κυρίως όσοι δεν είναι ευρωβουλευτές, ε, να καθίσουν, να είναι πιο ήσυχοι, να μπορέσουμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Και τώρα συγκεκριμένα Πρόκειται για τη συζήτηση για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, και θα θέλαμε να καλωσορίσουμε ε, δύο προσκεκλημένους που έχουμε, την κυρία Πέινς και την κυρία Τράουτμαν. Και τώρα θα ακολουθήσουμε την εξή διαδικασία. Κάθε μία εξ αυτών θα μιλήσει για περίπου 7 λεπτά και μετά θα έχουμε τη συνήθεια διαδικασία, πρώτα οι συντονιστές και μετά τα μέλη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα εδώ, δεν θέλω να χάσουμε χρόνο και θα ήθελα να δώσω το λόγο ε, και στις δυο σας. Η κυρία Πέις ίσως μπορεί να ξεκινήσει. Okay. Dear Chair, honorable members. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτά, κυρίες και κύριοι. Είμαι πανευτυχής γιατί είδα πώς ονομάστε την αίθουσα. Γιατί μιλούμε για έναν άνθρωπο που ήρθε για μένα πολιτικό ίνταλμα. Εγώ είμαι αρμόδια για το κεντρικό, ε, το διάδρομο κεντρικού δικτύου Ρήνου Δούναβη. Και σίγουρα είναι η ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, 6.000 χιλιόμετρα σιδηρόδρομου, 4.000 χιλιόμετρα οδικής ε, μεταφοράς και περίπου 9 ε, μέλη, πολλά χιλιόμετρα και εσωτερικών οδών ε, στο Δούναβι και το Σάβα. Και σίγουρα ο συντονιστή πρέπει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και πιστεύω με το επιτελείο μου καταφέραμε να πετύχουμε πολλά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως ε, θα σας εξηγήσω και στο έργο που ετοιμάζω, 96% του διαδρόμου έχει ε, ηλεκτροδοτηθεί και βέβαια υπάρχουν κάποια κενά σε κάποια διασυνοριακά σημεία, κυρίως μεταξύ Ουγγαρίας, Ρουμανίας, Γερμανίας και Τσεχίας και στη Ρουμανία. Σε ό,τι αφορά το ATMS, 7% είναι η συμμόρφωση στην Τσεχία Αυστρία και Ουγγαρία. Και σε ό,τι αφορά του εσωτερικού πλουτού 1% του διαδρόμου έχει ταξινομηθεί στην τέταρτη κατηγορία. Και σίγουρα χρειάζονται κάποιε βελτιώσει στη Γερμανία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και στην Κροατία κατά μήκο του ποταμού Σάβα. Και τα 80 ε, λιμάνια πληρούν τις προδιαγραφές του TNT για τις βασικές υποδομές η προμήθεια όμως για τα εναλλακτικά καύσιμα απέχει παρασάγκας από το στόχο. 80% σε ό,τι φέρει την οδική ασφάλεια είναι αυτοκινητόδρομοι, αλλά δυστυχώς ε, δεν έχουμε ε, διευθετήσει όλα τα, όλους τους στενοπούς και τα προβλήματα συμφόρησης. Το 2018 επισκέφθηκα το σημείο για τελευταία φορά. Έχουμε κάποια βελτίωση, αλλά θέλουμε να υλοποιήσουμε τους στόχους για την υλοποίηση του κεντρικού δικτύου μέχρι το 2030 έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μα. Από την έναρξη του συνδέοντο στην Ευρώπη το 2014, 101 ε, σχέδια ε, έχουν εφαρμοστεί, 3,5 δισεκατομμύρια το ύψος τους. Επίσης, Μέχρι στιγμής 3,07 δισεκατομμύρια είχαμε για τους ε, σιδηροδρόμους και 80% του συνολικού ποσού αφορούν τον διάδρομο. Για 141 παρεμβάσεις ε, που έχουμε τοπίσει στο πρόγραμμα εργασιών Μέχρι στιγμή 33 ε, έχουν υποστηριχθεί από το Μηχανισμό τη Ευρώπη και είμαι ιδιαίτερα περήφανη για τα αποτελέσματα τη Αιχία. Αντιμετωπίστηκαν οι στενοποί, Κυρίω ε, στο Μόναχο Νιρεβέργη Πράγα, σε αυτό το διάδρομο. Και έχουμε επιλύσει κάποιες στενοπού σε κάποια διασυνοριακά περάσματα. Αυτά τα σχέδια θα ολοκληρωθούν πλήρω μεταξύ 2020 και 2022 και εμπρόθεσμα μάλιστα. Στην Αυστρία και Γερμανία ε, πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σύραγγα στη Γερμανία. Ε, και σίγουρα χάρη στην ευληματική μας δράση για το Δούναβι έχουμε από τις 26 διαγωνισμούς δημόσιων συμβάσεων, 23 έχουν ολοκληρωθεί και περιμένουμε την παράδοση του εξοπλισμού. Επίσης, ολοκληρώνουμε περιβαλλοντικά προγράμματα στην Κροατία, Σλοβακία, Ουγγαρία και στο κοινό τομέα Βουλγαρίας-Ρουμανίας για να προετοιμάσουμε το μέλλον του δεύτερου μηχανισμού συνδέοντος Ευρώπη για τα οριζόντια θέματα. Η διαδικασία αναθεώρησης των κατευθυντήρων γραμμών του TNT έχει συνεχιστεί και θα πρέπει να δούμε και το, την καλή κατάσταση της ναυσιπλοείας. Θέλουμε καλή κατάσταση ναυσιπλοείας, GNS που λέμε, για τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Η έννοια αυτή της καλής κατάστασης ναυσιπλοείας αφορά το μέλλον της, των εσωτερικών πλωτών οδών. Γι' αυτό και έχουμε μια ειδική ομάδα εργασίας που θα συμβάλλει στην πρόταση για τον προσδιορισμό της καλή κατάστασης ναυσιπλοείας. Θα λάβουμε υπόψη φυσικά την πραγματικότητα των εσωτερικών πλωτών οδών και το ρόλο και την ε, ε, αρμοδιότητα των κρατών μελών, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή των εμπλεκομένων φορέων, των παρόχων υπηρεσιών και των διαχειριστών υποδομών. GNS σημαίνει μια καλή κατάσταση ναυσιπλοεία που θα εξασφαλίζει ασφαλή αξιόπιστη ναυσιπλοεία από του χρήστε με ε, εξασφάλιση ελάχιστων παραμέτρων και επιπέδων. Και η μελλοντική πολιτική μας για τις εσωτερικές πρώτες είναι πιο, πιο ελαστικές διατάξεις και κατάλληλες, ώστε να λαμβάνουμε υπόψη τα, διάφορα τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της εσωτερικής ναυσιπλοείας και να εξασφαλίσουμε εύρυθμη λειτουργία. Και μάλιστα θα υιοθετήσουμε προσέγγιση διαδρόμου για το καλή κατάσταση ναυσιπλοείας, ώστε να εξασφαλίσουμε την ε, ναυσιπλοεία αναδιάδρομο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ε, δεσμευθεί υπέρ ε, ενός βιώσιμου στήματος εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη. Όχι μόνο από τεχνική άποψη, ε, κάτι τέτοιο θα προωθήσει και τη συνοχή μεταξύ των χωρών. Για να ανταποκριθούμε όμως και να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις θα πρέπει να επιλύσουμε τα διάφορα σημεία. Σε ό,τι αφορά την ικανότητα απορρόφησης, το τμήμα συνοχή του διαδρόμου είναι κάτω από το κοινοτικό μεσόρο. 12 με 24 μήνες είναι καθυστερήσει ορευτικά. Ε, το συνδέεται στην Ευρώπη είναι ελαστικό μέσο, οπότε σε περίπτωση που δεν έχουμε αποδοτικά σχέδια, μειώνουμε τη συμμετοχή του στον προπολογισμό βέβαια. Ε, εξακολουθούμε να έχουμε κάποιους στενοπούς στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Θα πρέπει να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να θέσουν προτεραιότητα και να εθετήσουν έναν αγώ, όριμων σχεδίων, γιατί οι περισσότερες καθυστερήσεις οφείλονται σε προβλήματα στις δημόσιες συμβάσεις. Μερικές φορές και τέσσερα χρόνια κρατάνε οι διαγωνισμοί δημόσιων συμβάσεων. Συνήθως τέσσερα χρόνια χρειάζεται για την κατασκευή του έργου. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές κλίμα δημόσιων συμβάσεων για να ενισχύσουμε την αξιοπιστία των δημόσιων και ιδιωτών επενδυτών στις περισσότερες περιπτώσεις που έχουμε στεναπούς ε, είναι γιατί ένα κρατός μέλος από μόνο του δεν μπορεί να του αντιμετωπίσει. Θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τη συνεργασία, ιδιαίτερα όταν έχουμε εμπλοκή δύο-τριών κρατών μελών. Έχουμε επιτυχίες στο δικό μου διάδρομο, αλλά σίγουρα στις σιδηροδρόμους μεταξύ Γερμανίας και Τσεχίας και στις εσωτερικές πλωτές όδους μεταξύ Σερβίας και Κροατίας και Ουγγαρίας και Σλοβακίας θα πρέπει να εντείνουμε τι προσπάθειε. Θέλουμε μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική συνδρομή, όχι μόνο εθνικά, αλλά και σε επίπεδο διαδρόμου. Σας ευχαριστώ. Ähm, σας ευχαριστούμε πολύ ε, για την ε, εισήγησή σας σχετικά με το θέμα Ρήνος Δούναβης. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην ε, κυρία Τράουτμαν για την Βαλτική και την Ανατολική Θάλασσα. Ευχαριστώ. Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερος ε, που έρχομαι στην Επιτροπή Μεταφορών και βλέπω οικία πρόσωπα πρώην συναδέλφων ε, συμπεριλαμβανομένης και της Επιτρόπου. Τώρα, σήμερα θα λάβει χώρα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο η συζήτηση για τον προϋπολογισμό και θα είναι σημαντικό, όπως είπε και η Κάρλα Πέις, να λάβουμε υπόψη τους τρεις λόγους για τους οποίους θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ιδιαίτερα αυτό το διάδρομο Βόρειος Θάλασσας και Βαλτικής ε, που είναι σημαντικός για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ε, μεταφορών. Αυτός ο διάδρομος ε, είναι πολύ σημαντικός για την οικονομία. Έχουμε 12 θαλάσσιους λιμένες και μάλιστα από τους πιο σημαντικούς στο δυτικό τμήμα. Ρότερνταμ, Βέρσα για παράδειγμα, από τους σημαντικότερους λιμένες. Και σίγουρα αυτός ο διάδρομος είναι στρατηγικής σημασίας για την ασφάλεια και την άμυνα, γιατί συνδέει τις χώρες της Βαλτικής και περνάει από τη Βόρεια Θάλασσα στην Αρκτική Ζώνη, όπως ξέρετε, που επίσης αφισβητείται. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και πώς ε, θα την εφαρμόσουμε. Για μένα η κινητικότητα είναι από τις ε, σημαντικότερες δυνατότητες που έχουμε για να υλοποιήσουμε τους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια στιγμή που πρέπει να αποδείξουμε ότι θα εξασφαλίσουμε τα μέσα και τους πόρους για να έχουμε καλά αποτελέσματα και να μετριάσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες του δικτύου μου, του διαδρόμου μου και ε, τις βασικές προτεραιότητες που είναι η Via Baltica, Rail Baltica με τους, με τους σιδηροδρόμους που συνδέει το δυτικό με το ανατολικό τμήμα της Ευρώπης. Σημαντικός αυτή η σιδηροδρομική αρτηρία της Βαλτικής που δημιουργεί πολλές προκλήσεις και μας προβληματίζει. Θέλουμε ε, αποτελεσματικά σιδηροδρομικά δίκτυα με σημαντικές ταχύτητες μέχρι 250 χιλιόμετρα την ώρα μεταξύ Βαρσοβίας και Τάλιν και στις βαλτικές χώρες ήδη έχουμε εκτέλεση των ε, σχεδίων για 500 χιλιόμετρα από τα 870 χιλιόμετρα που έχουμε μέχρι στιγμής. Ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες προκατακτικές εργασίες και θα ακολουθήσουν και άλλες. Κάποιες αναβαθμίσεις ήδη γίνονται στην Πολωνία και θα έχουμε και μια νέα σιδηροδρομική γραμμή στο διοσυνοριακό τμήμα με τη Λιθουανία. Η βασική πρόκληση για την διαλειτουργικότητα των σιδηροδρόμων στο διάδρομό μου είναι να έχουμε ευρωπαϊκές προδιαγραφές και στη Βαλτική. Και γι' αυτό θα πρέπει να αναπτύξουμε το ERTMS. Γιατί ένα τμήμα μόνο του διαδρόμου είναι εξοπλισμένο. Θα πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τις επιδόσεις των σιδηροδρομικών μεταφορών και να συνδυάσουμε το μήκος με τη χωρητικότητα. Σίγουρα είναι από τους διαδρόμους με την υψηλότερη κυκλοφορία ναυτιλιακή. 27% του συνολικών εμπορευματικών μεταφορών που περνάνε από τα λιμάνια αυτά το 2018. Και σίγουρα και οι λιμένες ενδιαφέρονται για επαρκή σιδηροδρομική ικανότητα και συστήματα εφιών μεταφορών, προκειμένου να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα των ε, οδών πρόσβασης και στην εδωχώρα. Μερικοί λιμένες είναι ε, πρωτοπόροι σε θέματα ε, συστημάτων εφιών μεταφορών εναλλακτικών ε, καυσίμων και ψηφιοποίηση. Αλλά δυστυχώ αυτό είναι η εξαίρεση. Και υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι να αναπτύξουμε λύσει που δεν θα είναι τελικά διαλειτουργικές. Το 39% των επενδύσεων για τα προγράμματα αυτά στον ε, διάδρομό μου αφορούν κυρίως αστικού αστικούς κόμβους. Αν όμως δεν υλοποιήσουμε αυτά τα σχέδια θα έχουμε απώλεια 58 δισεκατομμύριων ευρώ σε ΑΕΠ και 220.000 ε, θέσεις απασχόλησης ε, θα χάνουμε το χρόνο την περίοδο 2015-2030. Βλέπετε στη δεύτερη διαφάνεια την πρόοδο που έχουμε σημειώσει στην εφαρμογή του διαδρόμου Βόρειας Θάλασσας και Βαλτικής. Μετά τις επενδύσεις στο διάδρομο έχουμε τον αριθμό των σχεδίων αναχώρα και βλέπετε ότι η Γερμανία έχει τα περισσότερα σχέδια. Η δεύτερη χώρα είναι η Πολωνία που επίσης συμμετέχει σε πολλά σχέδια, κυρίως στην επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου και βλέπετε και τις υπόλοιπες χώρες που επίσης εμπλέκονται ενεργά στην υλοποίηση των σχεδίων. 657 σχέδια έχουμε εντοπίσει συνολικά στο διάδρομο αυτό Βόρειας Θάλασσας και Βαλτικής, αξίας 110 δισεκατομμυρίων ευρώ επενδύσεων. Περίπου 35% των επενδύσεων αυτών έχουν σχέση ε, με σχέδια που συμβάλλουν άμεσα στα πρότυπα του κανονισμού ΤΕΝΤΗ και 23% των σχεδίων που είχαν συμπεριληφθεί στον κατάλογο από το 2014 ήδη έχουν διεκπαιρεωθεί. 65% αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2025. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπουμε τη, ε, τις επεκτάσεις του δικτύου από το 2021. Με τη θέση σε ισχύ του νέου κανονισμού για το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη, ο ε, διάδρομός θα επεκταθεί από το Ελσίνκι στο Λούλα της Σουηδίας, από το Βερολίνο στο λιμένα Στσέτσιν της Πολωνίας και από το Μαγδεβούργο στα σύνορα της Ουκρανίας μέσω του Κατοβίτσε. Θα είναι από τις σημαντικότερες επεκτάσεις ενός διαδρόμου, οι επεκτάσεις που σας αναφέρω από το 2021. Γιατί ο διάδρομος αυτός μας ενδιαφέρει και από στρατηγική άποψη, αλλά και άποψη πρώτων υλών. Θα πρέπει οπωσδήποτε να συνδέσουμε αυτό το τμήμα της Ευρώπης με το υπόλοιπο δίκτυο. Η επόμενη διαφάνεια αφορά τους διαδρόμους ως σημαντικούς παράγοντες διευκόλυνσης έξυπνων και βιώσιμων μεταφορών θέλουμε να κλείσουμε κενά και να καταργήσουμε στενοπούς σε ό,τι αφορά τις προσβάσεις στις αρτηρίες της Ευρώπης. Επίσης, συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων της Ευρωπαϊκής ε, Πράσινης Συμφωνίας με την ε, προσφορά υποδομών που χρειάζεται για τις ε, πολυτροπικές μεταφορές και τις αλυσίδε επιμελητίας και επίσης θέλουμε διαλειτουργικότητα με τις εσωτερικές πλωτές οδούς και σωστή διαχείριση των διαδρόμων που γίνεται με τη συμμετοχή των δημοσίων αρχών και των διαχειριστών των δικτύων σε όλα τα επίπεδα, τοπικό, περιφερειακό και εθνικό. Και παρά τη δημιουργία νέων φυσικών υποδομών, η πολιτική διευρωπαϊκών δικτύων στηρίζει και τις καινοτομίε, τις νέες τεχνολογίες και τις ψηφιακές λύσει, που θα πρέπει να καλύπτουν όλους τους τρόπους μεταφοράς. Η, η διάδρομη αυτή θα είναι η ραχοκοκαλιά για τη συνεχή ανάπτυξη διασυνοριακά ε, των ε, νέων σχεδίων. Και σίγουρα αυτή η προσέγγιση θα ενισχυθεί στην επικείμενη αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να αποφύγουμε τη, τα κενά ή τον κίνδυνο των κενών στο δίκτυο. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε και το φόρουμ για το Rail Baltica, γιατί θέλουμε να έχουμε συνδεδεμένες ε, υποδομές στην Ευρώπη. Θα γίνει στις 4 Μαρτίου του 2020 αυτό το φόρουμ για το σιδηροδρομικό Δίκαιο της Βαλτικής και σας προσκαλώ στο φόρουμ αυτό για να δείτε και η διεισόμαση σε ποια φάση του σχεδίου για το Rail Baltica βρισκόμαστε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Τρότμαν, κυρία Πέιν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις εισηγήσεις σας ε, και τώρα υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε συζήτηση. Ξεκινάμε λοιπόν με τους συντονιστές που είναι οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις. Οι συντονιστές έχουν καθίσει εξ αυτών τρία λεπτά στη διάθεσή τους. Ξεκινάμε με το ΕΛΚ και τη κυρία Τάλα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την εισήγησή σας, για την πολύ καλή δουλειά σας. Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για το δυναμικό, ανεκμετάλλευτο δυναμικό που υπάρχει στους σιδηρόδρομους. Ε, και γι' αυτό λοιπόν η ερώτηση μου αφορά ε, τους σιδηρόδρομους και απευθύνομαι και στις δυο σας. Βλέπετε να υπάρχει κάποιο είδος ε, ανταγωνισμού ανάμεσα στους συνδρομικούς φορείς που βρίσκονται στους διαδρόμους σας Μισό λεπτό. Ε, υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ με τη μετάφραση. Ε, Okay, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber äh, Συγγνώμη που σας ε, διακόψαμε. Είχαμε ένα μικρό τεχνικής φύσεως ε, πρόβλημα. Ε, ίσως μπορεί να ξεκινήσει και πάλι από την αρχή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ καλή δουλειά σας και την τις πολύ καλές εισηγήσεις. Όπως σας είπα ήδη, ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τους σιδηρόδρομους και για το πώς θα εκμεταλλευτούμε αυτό το ανακμετάλλευτο δυναμικό που υπάρχει στους σιδηρόδρομους. Γι' αυτό λοιπόν η ερώτηση μου αφορά τους σιδηρόδρομους και απευθύνομαι και στις δυο σας. Θεωρείτε ότι υπάρχει ίσως ε, κάποιος ανταγωνισμός ανάμεσα σε ε, σιδηροδρομικούς φορείς ε, που να βρίσκονται στους διαδρόμους σας και τι μέτρα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στους διαδρόμους. Ε, όγκο των εμπορευμάτων. Ποιο θα μπορούσε να είναι αυτός ο όγκο που να μεταφερθεί από, τους, από τις οδούς ε, στους σιδηρόδρομου, έχοντας πάντα κατά νου το σιδηροδρομικό δίκτυο. Και όσον αφορά την ε, μείωση της γραφειοκρατίας, ε, συνάδελφό σας Πατ Κόξ αναφέρεται σε low cost και no cost, δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει τι είδου μέτρα κρίνεται ότι είναι σημαντικά τα οποία θα μπορούσαν να αποδώσουν στους σιδηροδρόμους, ε, στους διαδρόμους σας και θα είναι και χαμηλού κόστους. Σάρφος από τους Σοσιαλδημοκράτες. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για τις δύο για τους ε, διαδρόμους όσον αφορά τον διάδρομο Ρήνου Δούναβη. Έχω δύο ερωτήσεις να υποβάλω, κυρίως όσον αφορά τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Ίσως μπορείτε να μας ε, πείτε περισσότερες λεπτομέρειες λεπτομέρειες για το ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, το αντιέξοδο που πρέπει να αντιμετωπιστεί στο Δούναβι για να διασφαλίσουμε καλή κατάσταση ναυσιπλοείας στο σύνολο της ε, εσωτερικής ε, πλωτής οδού. Και δεύτερον, τι ακριβώς χρειαζόμαστε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ε, αυξήσουμε για να πρασινίσουμε περισσότερο τις εσωτερικές πλωτές οδούς. Και μετά μία ερώτηση και προς τις δυο σας. Όσον αφορά τους σιδηρόδρομους, υπάρχει το, σύστημα των Ευρωπαϊκών, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Συνδρομικής Κυκλοφορίας. Εσείς ε, θεωρείτε ότι ε, μπορεί αυτό το σύστημα να επεκταθεί περαιτέρω στους δύο διαδρόμους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λυπάμαι πολύ. Πρέπει να φύγω τρέχοντας ε, από την ε, συνεδρία. Θα επανέλθω όμως, ε, εάν δεν προλάβω να ακούσω την ερώτηση, θα μου τη μεταφέρουν οι συνάδελφοί μου. Ευχαριστούμε πολύ, συνάδελφε, και επόμενος εκ μέρους της πολιτικής ομάδας Renew. Ο κύριος Ρικέ. Ευχαριστώ να χαιρετήσω τις δύο συντονίτριες. Εγώ θέλω να θέσω μια γενική ερώτηση στις δύο συντονίστριες. Καθώς ε, καταρχήν θέλω να ρωτήσω για το ρόλο που διαδραματίζεται και το δεύτερο είναι ότι έχουμε δύο διαδρόμους αρκετά διαφορετικούς από τεχνική σκοπιάς. Ε, θα ήθελα λοιπόν ε, να μου πείτε καθώς ε, ήδη εργάζεστε αρκετά χρόνια επί του θέματος, ε, σε, με ποια σειρά θα βάζετε τις δυσκολίες που σας εμποδίζουν να προχωρήσετε. Δηλαδή, βλέπουμε τέσσερα θέματα δυσκολίες Καταρχήν, δεν θα τα πω ε, με τη σειρά, εσείς να τα βάλετε στη σειρά από το πιο σημαντικό στο λιγότερο σημαντικό. Καταρχήν, έχουμε το οικονομικό κονδύλι. Δεύτερον, η δυναμία της τεχνικής ε, βοήθειας ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Τρίτον, πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών. Και τέταρτον, η διαφορά των πολιτικών επενδύσεων ε, μεταξύ των κρατών μελών και η δυσκολία για τα διασυνοριακά έργα. Επομένω, είναι περισσότερο τεχνικά, οικονομικά, πολιτικά. Τα προβλήματα ή σχετίζονται περισσότερο με τις συνδέσεις τις διασυνοριακές. Και έχω και δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Καταρχήν για το Ρήνο Δούναβι και το σχετικό διάδρομο, το GNS, στο δικό σας διάδρομο, Ρήνο Δούναβη. Πιστεύετε καλή κατάσταση ναυσιπλοεία. Πιστεύετε ότι μπορείτε να φτάσουμε στο 100% στο δικό σας διάδρομο και πιστεύετε ότι τα κλιματικά φαινόμενα και η λειψιδρία ή μάλλον αν έχουμε χαμηλή στάθμη μπορεί αυτό να έχει αντίκτυπο στη συνέχιση της υλοποίησης του ποτάμιου διαδρόμου. Και σε ό,τι αφορά τώρα Βαλτική Βόρεια Θάλασσα και το σχετικό διάδρομο, μπορείτε να μας πείτε τις δυσκολίες ε, με περισσότερες λεπτομέρειες μέσα σε εισαγωγικά αυτό για τις ε, διασυνοριακές ή τις διακρατικές ε, δομές για το Transbaltica. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ και επόμενος η επόμενη εκ μέρους των Πρασίνων, ε, συνάδελφος ε, Ντεπανέ. Πολύ σωστά προφέρατε ε, το όνομά μου, λέγομαι Ντεπανέ Γκρούνεμπερκ. Κατ' ουσίαν όταν προφέρει κανείς το όνομά μου είναι σαν να κάνει εξάσκηση στα αγγλικά και στα, γερμανικά, στα γαλλικά και στα γερμανικά. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα αυτά που μας είπατε και ευθύ εξ αρχή να σας πω ότι η κινητικότητα βεβαίως είναι η σπονδυλική στήλη της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Γι' αυτό λοιπόν το να ασχοληθείτε με αυτό αυτούς τους διαδρόμους. Είναι ε, πάρα πολύ σημαντικό για μας. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σας. Και επειδή έχουμε ένα αντιμετωπίσουμε δύο νέες μεγάλες προτεραιότητες με την Επιτροπή. Έχουμε να υλοποιήσουμε το πρασίνισμα, την μείωση των εκπομπών, την κρίση της βιοποικιλότητας. Απευθύνομαι και στους δυο σας. Ε, τελικά έχετε νέες προτεραιότητες. Δηλαδή, ε, μερικές φορές ε, ισχύει ή προσπαθούμε να αναθεωρήσουμε τα προγράμματα και να εφαρμόσουμε νέα κριτήρια. Και θα ήθελα να αναφέρω και κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα και ερωτήσεις. Στο μέλλον πώς θα αξιολογούμε τα μεγάλα προγράμματα. Ε, σε αυτό το διάδρομο ε, Ρήνου ε, Δουνάβεως είχαμε το πρόγραμμα Στουτγάρδη 21. Εγώ έρχομαι του Στουτγάρδη και εκεί υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε 28 εκατομμύρια για ένα project το οποίο συνολικά τελικά θα κοστίσει πάνω από 8 δισεκατομμύρια. Εσείς τι λέτε, αυτά τα χρήματα δαπανήθηκαν σωστά τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν καθοδόν ε, διάφορες αδυναμίες, μικρά, κενά, ε, ως εκ τούτου θα πρέπει στο μέλλον να επανεξετάσουμε τις προτεραιότητές μας. Και την ερώτηση μου τη συνδέω με αυτό που ρώτησε ο κύριος Ρικέ. Δηλαδή, ποια είναι ε, τα επενδυτικά, τα προβλήματα που μας ε, συνοδεύουν. Είναι επενδυτικά, είναι διοικητικά. Πού ακριβώς πρέπει να επενδύουμε. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα κατά νου. Ε, παρεμφερεί τα προβλήματα και με, με την Πράσινη Συμφωνία. Προάγουμε δηλαδή ε, προγράμματα όπου βλέπουμε ότι υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα τις οδικές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Έχω κατά νου κυρίως τη Βαβαρία και την Τσεχία. Και τι είδαμε, ότι οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι αποφάσισαν να εγκαταλείψουν σιγά σιγά τους σιδηρόδρομους και να μεταφέρουν τους επιβάτες περισσότερο με λεωφορεία. Άρα δηλαδή αυτό είναι πρόβλημα. Είναι όμως πρόβλημα και για τις εμπορευματικές μεταφορές και για τα βραδινά δρομολόγια. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας ερωτήσω τι σκέπτεστε να κάνετε. Και έχω και δύο προβλήματα που θέλω να θίξω καταλήξω σε σχέση με την βιοπικιλότητα, ε, κυρία Πάγες. Ε, καταρχήν, ε, όσον αφορά την ναυσιπλοεία στο Δούναβι, στο πώς καταστρέφεται το οικοσύστημα στο Δούναβι και τι θα γίνει εφαρμοστούν τα προγράμματα που παρουσιάσατε. Κυρία Τράουτμαν, προς εσάς έχω μία ερώτηση σε σχέση με τη βιοπικιλότητα. Στην παραμεθόρια περιοχή, ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λιθουανία, έχουμε παρθένα δάση, ε, πραγματικούς ε, θησαυρού με μεγάλη βιοπικιλότητα. Και ε, ίσως εκεί θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το τι θα κάνουμε με τους διαδρόμους, διότι όπως ακούσαμε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει νέε προτεραιότητε. Σα ευχαριστούμε πολύ για τη δουλειά σα και καλό κουράγιο και για τη συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμεί, ε, λέει ο πρόεδρο. ID, ECR και GUE ε, ε, δεν έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να ερωτήσουν μέσω συντονιστών. Γι' αυτό λοιπόν θα έλεγα τώρα να ακολουθήσουν οι βουλευτές εφόσον θέλουν να κάνουν ερωτήσεις και στο τέλος να δοθούν οι απαντήσεις. Επόμενη συνάδελφος είναι η συνάδελφος Τεξ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ε, θα μιλήσω Ολλανδικά. Κυρίως για να δώσω το αίσθημα στην κυρία Πέις ότι είναι στο σπίτι της. Εγώ έρχομαι από το Φένλο και εκεί οι πολίτες μου λένε ότι ενδεχομένως ε, να υπάρξει πρόβλημα εάν τα κονδύλια από τη διευκόλυνση συνδέοντας Ευρώπη δοθούν ε, το 20, αλλά τα επόμενα για τα 5T το 21 με αυτή τη χρονική διαφορά. Κατ' ουσίαν τι σημαίνουν όλα αυτά. Το πρώτο χρονικό διάστημα ε, όπου θα εφαρμόζεται το, ο μηχανισμός διευκόνησης Ευρώπης, κατά το πρώτο ήδη χρονικό διάστημα θα έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια. Όσοι μετά θα ακολουθήσουν δεν θα επωφεληθούν. Επ' αυτού το έχετε λιγάκι σκεφτεί. Έχετε σκεφτεί τι είδου λύση θα μπορούσε να βρεθεί σε αυτό το θέμα. Πολύ ωραία. Επόμενος, ε, συνάδελφος Μπέρενσον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τις δυο σας ε, για όλα αυτά που μας είπατε. Η δική μου ερώτηση έχει σχέση περισσότερο με το ρόλο σας ως ε, Ευρωπαίοι συντονιστές. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο ε, για τον e, ΕΦΗ φάκελο τεντή, γιατί για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ε, κυρίως οι διασυνοριακές, δηλαδή τα χρονοδιαγράμματα, οι αδειοδοτήσεις. Επίσης, ε, εξετάζουμε το ρόλο και των Ευρωπαίων συντονιστών. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω από εσάς αυτή τη στιγμή ποιο είναι το όραμά σας με βάση τα εργαλεία που έχετε στα χέρια σας. Και επίσης, πώς θα να ενισχυθεί η θέση σας έχοντας πάντα κατά νου την αρχή της επικουρικότητας. Να ε, επιταχυνθούν οι διαδικασίες κυρίως όταν πρόκειται για ε, διασυνοριακά προγράμματα. Συνάδελφος Γκίζεκε, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και τι δύο εισηγήτριε. Ε, η Πράσινη Συμφωνία αυτή τη στιγμή είναι το βασικότερο θέμα. Και νομίζω ότι η ολοκλήρωση των ε, διαδρόμων αυτών μπορεί να συμβάλλει για να επιτύχουμε του στόχου τη πράσινη συμφωνία. Βέβαια, μπορούμε να διορτηθούμε Πώ θα τα καταφέρουμε όλα αυτά ακούει, ακούσει κανείς αυτά που είπατε κυρία Πέις, θα καταλήξει συμπέρασμα ότι η διαδικασία ανάθεσης έργων αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη διαρκεί τέσσερα χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Ε, θα πρέπει να αναλυφθούν πρωτοβουλίες για να υπάρχει επιτάχυνση. Υπάρχει και μια πρωτοβουλία του κυρίου Σεύκοβιτς ε, που έχει στόχο την επιτάχυνση των προγραμμάτων. Μπορούμε λοιπόν ίσως να μεριμνήσουμε ώστε οι διαδικασίες εφαρμογής να επιταχυνθούν και τέλος κάτι που έχει σχέση με τα κονδύλια. Αυτή τη στιγμή οι δημοσιονομικές διαπραγματεύσεις ε, τρομάζουν λιγάκι γιατί από ό,τι φαίνεται ε, απομακρυνόμεθα από το στόχο του ε, Κοινοβουλίου 1,3 του ΑΕΠ. Τα κράτη-μέλη είναι πολύ πιο συγκρατημένα. Γι' αυτό και τα κράτη-μέλη πρέπει να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή των διευρωπαϊκών δικτύων TNT. Πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Και έχω και μία τεχνική ερώτηση. Αναφερθήκατε στην καλή κατάσταση τη ναυσιπλοεία, κυρία Πέη. Το 2005 όσον αφορούσε τις εσωτερικές πιλωτές οδούς είχαμε το River Information System Τώρα έχουν περάσει πέντε χρόνια, πρέπει να το αναθεωρήσουμε. Ίσως πρέπει να επικαιροποιηθεί το σύστημα αυτό. Ε, και στην κυρία Τράουτμαν, όσον αφορά τη Rail Baltica, το 2023 ε, υποτίθεται είναι καταληκτική ημερομηνία. Θα τα καταφέρουμε. Αυτά τα joint ventures, οι κοινοπραξίες, είναι μια σωστή δομή για να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2023. Κατά τα άλλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή δουλειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κίζικε. Επόμενος συνάδελφος Νταλούντε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα θέσω κάποιες ερωτήσεις ε, σε ό,τι αφορά το θέμα της διακυβέρνησης, το governance. Υπάρχει μια μακρά ιστορία που μιλά για έλεγχο της συνδρομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ε, ε, στις υποδομές, τις απανομές των χρονοθυρίδων, τις τιμές ε, των τρένων και γι' αυτό πιστεύουμε ότι ένας καλύτερος συντονισμός θα έπρεπε να μην βασίζεται σε εθνική αλλά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τι άλλα ε, πολιτικά ε, ποιο άλλο πολιτικό βάρος χρειάζεστε, πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε εμείς, ποια άλλα εργαλεία και μέσα μπορούμε να θέσουμε στα χέρια των συντονιστών για να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή διακυβέρνηση ακόμα και μέσω του Ευρωπαϊκού ε, Σιδηροδρομικού Οργανισμού Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ένα καλύτερο ευρωπαϊκό σχεδιασμό σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις, τι υποδομές, ε, τη διαχείριση των χρονοθυρίων, την τιμολόγηση κτλ. Τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε εμείς, ε, λοιπόν, για να έχουμε καλύτερη διαχείριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. von der EVP, die Kollegin Hanna thank you, Mr. Κυρία Βερκουνέν, σας ευχαριστώ. Μιλάμε τώρα για πολύ σημαντικά ευρωπαϊκά δίκτυα. Ξέρουμε ότι είναι ζωτικά για την ανταγωνιστικότητα, για την ενίαγορά αγορά και για να μειώσουμε τις ε, εκπομπές άνθρακα στις μεταφορές. Σήμερα έχουμε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα συζητήσει τον πολιτή προπολογισμό μας ε, και δεν είμαι πολύ αισιόδοξη γιατί προτείνουν ε, μεγάλες περικοπές στο μηχανισμό ΣΕΦ και ε, έχουμε πάρα πολλές περικοπές ε, ζωτικές για τα έργα. Θα ήθελα να μας πείτε εσείς πόσο θετικές είστε για την εφαρμογή των έργων, πώς το βλέπετε και πώς ρώτησαν πολλοί συνάδελφοι, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις, είναι το θέμα της χρηματοδότησης. Επίση, ακούσαμε ότι σε ορισμένε χώρες τα κράτη-μέλη έχουν ε, πρόβλημα σε σχέση με το να θέσουν τα έργα σε προτεραιότητα και οι διαδικασίες προμηθειών είναι πολύ αργέ σε κάποια κράτη-μέλη. Ποιες είναι οι κύριε προκλήσεις, ε, λοιπόν, κατά τη γνώμη σας για την εφαρμογή των διαδρόμων ή την υλοποίηση των διαδρόμων. Ο κύριο Νταλούντε επίση αναφέρθηκε στο πώ μπορούμε να υποστηρίξουμε το δικό σα έργο για να μπορούμε να υλοποιήσουμε τους διαδρόμους. Η αναθεώρηση των μεταφορών είναι τώρα υπό εξέλιξη και φυσικά θα υπάρχουν κάποιες επεκτάσεις στο διαδρόμο. Εγώ προέρχομαι από τη Φιλανδία και φυσικά είμαστε ικανοποιημένοι που τώρα έχουμε στο χάρτη και την επέκταση στη Σκανδιναβία γιατί πριν η Σκανδιναβία δεν ήταν ιδιαίτερα στο χάρτη των μεταφορών. Όμως υπάρχουν και άλλα στοιχεία που βλέπετε ότι θα πρέπει να προσθεθούν σε αυτούς τους διαδρόμους ε, τώρα που αναφερούμε το δίκτυο ΔΕΔ, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Τελευταίο ε, ερωτών στον κατάλογό μου είναι ο συνάδελφος Σαλίνη από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ήμουν σε μια συζήτηση σε μια άλλη επιτροπή που αφορά το θέμα των ασφαλιστικών δικλείδων στη βιομηχανία. Εντυπωσιάστηκα γιατί κατά διάρκεια της συζήτησης ε, είχαμε, λάβαμε ένα ακαδημαϊκό μάθημα από την Κομισιόν ε, και μας εξήγησε με πάσα λεπτομέρεια το πώς πρέπει να ερμηνεύονται οι κανόνες ε, για να ε, έχουμε μία τέλεια ερμηλεία του δόγματος του ΠΟΕ. Και εδώ θέλω να σημειώσω ότι ίσως κάποιος δεν αντιλαμβάνεται ότι στην Ιταλία ο κλάδος, η βιομηχανία χάνει και στην Ευρώπη χάνει σε ανταγωνιστικότητα, σε θέσεις εργασίας, δυσκολευόμαστε να έχουμε παρουσία στις παγκόσμιες αγορές πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Επομένως, καθώς βρισκόμαστε ενώπιον μιας ε, σημαντικής ε, ε, επίγουσας οικονομικής κατάστασης, δεν νομίζω ότι ο κύριος ε, στόχος μας σήμερα είναι να μιλάμε μόνο για τον Πράσινη Συμφωνία, αλλά να μιλήσουμε για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια αγορά. Και καθώς ε, αναθεωρούμε τον κανονισμό για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τουλάχιστον μερικώς, ε, κάνω το ακόλουθο αίτημα. Εμείς πρέπει να καταλάβουμε αν μπορούμε να είμαστε φιλόδοξοι. Φιλόδοξοι. Η συζήτηση για τον προπολογισμό αυτή τη στιγμή δεν είναι φιλόδοξη και παίρνοντα χάρη τα κονδύλια που έχουμε για το ΣΕΦ δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά. Φαίνεται ότι υπάρχουν εσωτερικέ δυνάμει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε που θέλουν ουσιαστικά να κάνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να υπαναχωρήσει. Επομένω, για αυτή την αναθεώρηση των κανόνων για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, θέλουμε η πολιτική συζήτηση να είναι φιλόδοξη προκειμένου στου ευρωπαϊκού λαού να προσδώσουμε εμπιστοσύνη είναι ότι εμείς θα προωθήσουμε την ανάπτυξη υλοποιώντας μέσω μαζικών επενδύσεων στις υποδομές αυτό που θέλει ο πληθυσμός. Ανάπτυξη δηλαδή, όχι θεωρητικές συζητήσεις. Vielen ähm, Es gibt keine weiteren Fragen von den Abgeordneten ich würde Ihnen... Δεν έχουμε άλλε ερωτήσει από τους βουλευτές και θα ήθελα τώρα να δώσω τη δυνατότητα και στις δυο σα να τοποθετηθείτε ε, σε αυτά τα οποία ε, ερώτησαν οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο Uh, competition in my... Λοιπόν, για τον ανταγωνισμό στο δικό μου διάδρομο και πόσο από τα εμπορεύματα μπορούν να πάνε στο Ρήνο. Θεωρητικά τα πάντα. Αλλά χρειαζόμαστε, συγγνώμη, μπορώ να πάνε σε μεταφορέ, αλλά χρειάζεστε σιδηροδρόμου ε, πρώτα. Και κατόπιν θα φτάσω στι ε, διαδικασίε ε, που οδηγούν στι καθυστερήσει που έχουμε αλλά δεν νομίζω ότι ο ανταγωνισμό είναι η μεγαλύτερη ανησυχία στι χώρε συνοχή. Έξι χώρε συνοχή είναι στο δικό μου διάδρομο. Ο ανταγωνισμό δεν είναι η πρώτη μου ανησυχία. Η πρώτη μου ανησυχία είναι σιδηρόδρομη και πιθανότατα με το ERTMS και την δυνατότητα των ανθρώπων να πάνε από το Α στο Β και νομίζω ότι είναι αυτό το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή και κατόπιν έχουμε πολλές εταιρείες ε, που μπορείς να, μπορείς να ακολουθήσεις αυτήν την κατεύθυνση, αλλά καταρχήν χρειαζόμαστε τις ίδιες τις υποδομές. Μετά είχαμε την ερώτηση του κυρίου Ντάνιελσον. Ποια είναι η κύρια εμπλοκή. Λοιπόν, από το Στρασβούρο στην Κωνσταντσα, αν θες να πας εκεί, έχουμε δύο σημεία προβληματικά. Καταρχήν έχουμε το θέμα του κλίματος, ε, γιατί ε, εμείς ε, δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Εξακολουθούμε να έχουμε περίοδο χαμηλή στάθμης του νερού, όχι μόνο στο Δούναβι, το καλοκαίρι, αλλά και στο Ρήνο. Το κλίμα είναι πραγματικά πρόβλημα και πρέπει να ζήσουμε με αυτό. Μπορούμε να κάνουμε το οτιδήποτε, αλλά ε, δεν ε, ξέρω αν μπορούμε να ελέγξουμε το επίπεδο του νερού. Ε, αυτή τη στιγμή να το λύσουμε ολοκληρωτικά δεν μπορούμε. Επίσης έχουμε το, προ... το project Strobik Vilsov και δεν ε, είναι δυνατόν στο μέλλον να χρησιμοποιήσουμε πλήρως ε, τις συνδέσεις ε, μεταξύ του Ρήνου και του Δούναβη. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι σε κάποιες από τις χώρες συνοχής έχουμε πολιτική αστάθεια. Είναι αδύνατο ένα συντονιστή να πάει σε μια χώρα που δεν υπάρχει υπουργό γιατί οι αρχέ ε, πρέπει να ξέρουν ότι βρίσκομαι στη χώρα και τι κάνω εκεί και πολλέ φορέ ε, θέλω να μιλήσω με τι αρχέ. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Λοιπόν, ε, αυτά είναι τα πιο σημαντικά προβλήματα. Στι διαδικασίε θα αναφερθώ αργότερα. Εναλλακτικά καύσιμα. Είναι πραγματική πρόκληση. Και όχι μόνο γιατί κανείς δεν θέλει να επενδύσει στα εναλλακτικά καύσιμα, αλλά χρειάζεσαι επίσης και αρκετά πλοία, χρειάζεσαι πελάτες. Ε, αν έχεις μια ολόκληρη λυσίδα εναλλακτικών καυσίμων, χρειάζεσαι και πλοία που να έρθουν να αγοράσουν αυτά τα καύσιμα. Αλλά κανείς δεν επενδύει. Όλα αυτά είναι αλληλοσυνδεδεμένα. Αν επιλύσουμε το θέμα της υποδομής θα έρθουν και εναλλακτικά καύσιμα. Υπάρχουν κονδύλια, δεν είναι πρόβλημα αυτό. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε το ERTMS, το σύστημα διαχείρισης του Και στη δική μου χώρα το ERTMS κάνει πολύ πιο ασφαλή και πιο γρήγορη την υποδομή. Μπορείς να έχεις περισσότερα σε μία σιδηροδρομική γραμμή. Είναι ακριβό, αλλά αποπληρώνει. Και μόλις το δουν οι άνθρωποι, νομίζω ότι θα βελτιώσουν το ERTMS. Κυρίως ε, σε τροχές που χρησιμοποιούνται πάρα πολύ. Κύριε Ρικέ, είπατε κάτι για θέσπιση προτεραιοτήτων αλλά τι είπατε εμένα, ρωτήσατε ή τη συνάδελφο, την κυρία μου Και τις δύο. Και στις δύο α, απέφθηνε την ερώτησή μου. Ποιες θεωρείτε ότι είναι μεγαλύτερες δυσκολίες σας. Είναι δημοσιονομικές, χρηματοδοτικές, δηλαδή διοικητικές ή πολιτικές. Χωρίς μικρόφωνο, κυρία Πέις. Είναι πάσης φύσεως τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρεί ένα σχέδιο. για να επιλέγετε ή να αποκλείετε. Φυσικά θα πρέπει να κάνουμε μία επιλογή, να έχουμε προτεραιότητες γιατί δεν υπάρχουν πολλά κονδύλια δεν είναι απεριόριστα. Θα πρέπει λοιπόν να καθορίσουμε τις προτεραιότητές μας και να χρηματοδοτούμε τα σχέδια ύψης της προτεραιότητας. Η χρηματοδότηση ποτέ δεν είναι επαρκής. Δεν είναι ανεξάντλητη η πόρη και τα κονδύλια μας, αλλά αυτό το γνωρίζουμε. Τώρα, οι διαδικασίες, επίσης σημαντικό θέμα. Γιατί αν δούμε τους διαγωνισμούς στις δημόσιες συμβάσεις, το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε μια νέα διαδικασία για τους διαγωνισμούς. Πέραν τούτου όμως, ε, και δεδομένου ότι πρέπει να απλουστεύσουμε την γραφειοκρατία, ε, βλέπουμε ότι παρόλα αυτά υπάρχει τέτοιο χαρτομάνι, τέτοιες γραφειοκρατικές διατυπώσεις που μερικές χώρες ε, έχουν καθυστερήσει δύο και τέσσερα χρόνια. Και διαρωτόμαστε αν θα μπορούσαμε να επιταχύρουμε τη διαδικασία των διαγωνισμών. Το συζητήσαμε με όλες τις χώρες και είπαμε ότι θα βρούμε κάποιες λύσεις. Μερικές χώρες τις βρήκαν μόνες τους τις λύσεις να επιταχύνουν τις διαδικασίες και να καταλήξουν ταχύτερα σε συμφωνία με τον ανάδοχο. Συγγνώμη, μακρηγόρησα. Θέλουν να, να επιταχύνουν τις διαδικασίες και τις προθεσμίες στον διαγωνισμό. έτσι μπορούμε να κερδίσουμε και δύο χρόνια που είναι καταπληκτικό επίτευγμα αν επισπεύσουμε κατά δύο χρόνια τους διαγωνισμούς. Και μάλλον οι δημόσιες διατάξεις στην επόμενη φάση τουλάχιστον δεν θα είναι το μείζον πρόβλημα. Είχα πολλές ερωτήσεις. Τι να κάνω, δεν προλάβαινα πιο γρήγορα. Η κυρία Τροτμάν. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γαλλικά τώρα για να συγκεντρώσω τις απαντήσεις μου σε συγκεκριμένα θέματα. Καταρχήν για τους σιδηροδρόμους. Σε αυτή τη φάση περιμένω να αποδώσουμε την ίδια σημασία στις εμπορευματικές μεταφορές σιδηροδρόμων και στις μεταφορές επιβατών τις σιδηροδρομικές. Επίσης, να επιταχύνουμε την ε, μεταφορά και των φορτηγών με σιδηροδρομικές μεταφορές. Πριν από λίγες μέρες ένα τρένο ξεκίνησε από το Βεταμβούρ για το Πόσναν. Είναι μεταφορά μεγάλης απόστασης, αλλά θα μπορούσαμε να ενώσουμε λιμάνια ή πλατφόρμες εμπορευματικών μεταφορών στα διάφορα σημεία της Ευρώπης. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Τρίτον, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις ε, πλατφόρμες της επιμελητίας, γιατί μιλούμε για υποδομές, αλλά ας μιλήσουμε και για ροές, για οικονομίες, για οικονομικά κέρδη, γιατί όσο πιο γρήγορα ολοκληρώσουμε τις υποδομές, τόσο πιο γρήγορα θα δρέψουμε τους καρπούς και τους οικονομικούς. Και σίγουρα τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών είναι επιταχυντής και σε ενεργειακά και σε οικονομικά θέματα. Με τη δέσμευση άνθρακα, για παράδειγμα, αλλά είναι και οικονομικό επιταχυντή. Αυτό το διαπιστώνουμε στο δικό μου διάδρομο Βόρεια Θάλασσα και Βαλτική. Γιατί από την αρχή θεωρήσαμε αυτό το διάδρομο ω οικονομικό διάδρομο, κινητοποιώντα επιχειρήσει, διευκολύνοντα την προσέλκυση και επενδυτών ή και των λιμένων σε διάφορα μέρη. Το λιμάνι του Αμβούργου επένδυσε στο Τάλιν. Οι κάτω χώρες με το Ρότερνταμ κάλυψαν το σύνολο του διαδρόμου. Θέλουμε ο διάδρομος αυτός ε, να χαρακτηριστεί από μια οικονομική ολοκλήρωση και αυτό θα είναι το μείζον κέρδος και επίτευγμά μας. Επίσης, οφείλουμε να έχουμε μια στρατηγική επιτάχυνσης. Έτσι θα βελτιώσουμε και τον ανταγωνισμό, αλλά ταυτόχρονα θα πραγματοποιήσουμε εκ παραλίλου διάφορα έργα. Για παράδειγμα, στον διάδρομό μου για το Rail Baltica ταυτόχρονα κατασκευάζουμε και γέφυρες. Συγκεκριμένο παράδειγμα που μας επιτρέπει να τηρήσουμε τις προθεσμίες και να επιταχύνουμε τη διεκπαιρέωση. Και είναι σημαντικό αυτό για την αξιοπιστία μας απέναντι στους πολίτες και για να δείξουμε και εμπράκτος ότι η πολιτική μεταφορών είναι χρήσιμη από κάθε άποψη. Επίσης, στο θέμα των προτεραιοτήτων. Σήμερα έχουμε το πρόβλημα της χρηματοδότησης, αλλά έχουμε ταυτόχρονα και το επίπεδο των κονδυλίων και των επιδοτήσεων, αλλά και η δημοσιονομική βιωσιμότητα, αν θέλουμε να συνδυάσουμε τις διάφορες πηγές χρηματοδότησης. Και γνωρίζουμε επίσης πόσο ανάγκη έχουμε αυτό το συνδυασμό. Και η δημοσιονομική η χρηματοδοτική βιωσιμότητα αφορά την βιωσιμότητα και των αποφάσεών μας και τη δυνατότητα του να έχουμε το ίδιο επίπεδο χρηματοδότηση καθ' όλη τη διάρκεια της υλοποίηση του σχεδίου και εμπροκειμένου μέχρι το 2030. Και αυτό δεν έχει ληφθεί δεόντω υπόψη στη συζήτηση που γίνεται. Γιατί μειώνεται το κονδύλιο για την ε, στρατιωτική κινητικότητα και μειώνουμε δυστυχώς και το μηχανισμό συνδέοντας στην Ευρώπη. Θα πρέπει για τα μεγαλοεπίβολα σχέδια να βρούμε και την κατάλληλη διακυβέρνηση. Το βλέπω για το Rail Baltica, καλό παράδειγμα και η μεγαλύτερη δυσκολία του είναι ότι μερικές χώρες θεωρούν αυτή την υποδομή ως εθνική υποδομή και ως τμήμα δηλαδή και όχι ως σύνολο. Εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε τους, μπορείτε να βοηθήσετε τους συντονιστές επιμένοντας στην ε, προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία που έχουν όλα αυτά τα σχέδια σε ό,τι αφορά την βιοπικιλότητα. Σίγουρα μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας υπάρχουν κάποιες υγρές ζώνες ε, παρθένων δασών και αρχαίγωνων δασών ε, πολύτιμες για τη βιοπικιλότητα και λαμβάνονται υπόψη οι ζώνες αυτές. Στην Πολωνία έχουμε μια επιστημονική επιτροπή που απεφάνθη υπέρ της πραγματοποίησης ε, αυτής της υποδομής, της κατασκευής αυτής της υποδομής. Φυσικά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την προστασία της χλωρίδας και πανίδας τοπικά και προχωρούμε στο δίκτυο ταυτόχρονα με τα επιστημονικά πορίσματα και την περιβαλλοντική αξιολόγηση αντικτύπου. Επίσης, ό,τι αφορά τους συντονιστές, τι θα μπορούσατε εσείς να κάνετε για να βοηθήσετε τους συντονιστές. Ίσως να μεταφέρετε, να διαβάσετε τα αποτελέσματά μας, γιατί Σήμερα ίσω θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με του υπουργού και του αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων, γιατί εκείνοι έχουν στα χέρια του το, το γκάζι. Εκείνοι μπορούν να επιτυχύνουν την κατάσταση. Βέβαια, τα νομοθετικά αισθήματα δεν είναι τα ίδια παντού. Και σίγουρα έχουμε πρόβλημα συντονισμού. Και για το Rail Baltica είδαμε καλό συντονισμό των βουλευτών με τη λέσχη φίλων του σιδηροδρόμου της Βαλτικής. Εκεί πραγματικά είχαμε μία επιτάχυνση με πολύ θετική επιρροή των βουλευτών. Θα πρέπει λοιπόν και να μεταφέρετε προς τα έξω τα αποτέλεσματά μας και να συνεργάζεστε μεταξύ και με τις κυβερνήσεις σας για να προωθείτε και να επιταχύνετε τα διάφορα σχέδια. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε την κυρία Πέις και την ε, κυρία Τροτμάν για τις απαντήσεις τους και σας ζητώ συγγνώμη που χρειάζεται και να σας επιβάλλω ε, μια αυστηρότητα χρόνου αλλά δεν έχουμε χρόνο. Δύο λεπτά ακόμη και μετά θα πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μιλήσατε για τις νέες προτεραιότητες. Φυσικά η Ευρωπαϊκή Νέα Πράσινη Συμφωνία είναι τεράστια προτεραιότητα και αναπόφευκτη για την επόμενη περίοδο. Και αυτό θα είναι σημαντικότατη πρόκληση. Στουτκάρδη. Θα ήθελα να πω το εξής για τη Στουτκάρδη. Δεν πληρώσαμε για το σταθμό. Μόνο για τις γραμμές, τις ράγες. Τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει το κράτος μέλος και η πόλη, ο Δήμος. Εμείς μόνο τις γραμμές τις σιδηροδρομικές ε, χρηματοδοτήσαμε γιατί πρόκειται για αστικό κόμβο και γι' αυτό επενδύσαμε εκεί στη Στουτκάρδη. Τώρα αν υπάρχει πρόβλημα μεταξύ Μονάχου και Πράγας μεταξύ σιδεροδρομικών και οδικών μεταφορών. Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αντίθετα, επιταχύνουμε τα πράγματα εκεί και πάνε μια χαρά. Η γερμανική κυβέρνηση μας βοήθησε πολύ στο να μπει αυτό το σχέδιο στο κατάλογο των σχεδίων υπό υλοποίηση. Τώρα, η, ο αντίκτυπος στην αυσιπλοεία του Δούναβη. Φυσικά θα υπάρξει ε, επιρροή της ναυσιπλοείας στο Δούναβι, αλλά υπάρχει και επιρροή των φορτηγών και των μεταφορών με φορτηγά στο περιβάλλον. Και σίγουρα η ναυσιπλοεία έχει λιγότερο επιζήμιες περιβαλλοντικές συνέπειες από ε, τις οδικές μεταφορές ή τις εναέρειες μεταφορές. Κυρία Τάξη. Τώρα για το υπόλοιπο θέμα που ρωτήσατε θα πρέπει να το εξετάσω. Δεν έχω ιδέα, είμαι απροετοίμαστη. Πάντως δεν έχουμε αρμοδιότητα για τον σημερινό προπολογισμό και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των δημοσιονομικών διαπραγματεύσεων. Ο ρόλος των συντονιστών τώρα και πώς μπορούμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, ιδιαίτερα για διασυνοριακά σχέδια. Αυτό είναι όντως πρόβλημα και εμείς ως συντονιστές οι συντονίστρες θα πρέπει να συμμετέχουμε. Το είδαμε στην περίπτωση Βουλγαρίας και Ρουμανίας ότι είναι καλύτερο να συμμετέχουμε γιατί έτσι μπορούμε να προωθήσουμε και τα πράγματα. Και έτσι έχουμε το πρόγραμμα για την συνεργασία στον κοινό τομέα Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Κύριε Φάλκα, πρασίνισμα και δημόσιες συμβάσεις για το συνδέοντα στην Ευρώπη. Φυσικά θα επενδύουμε σε αυτά τα θέματα. Είναι υποχρέωσή μας και καθήκον μας. Σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και για τις απαντήσεις που μας δώσατε. Νομίζω ότι καλύψατε όλα τα θέματα. Το γνωρίζω, ε, λέει κυρία γιατί ήμουν για 14 χρόνια ευρωβουλευτής. Ξέρω ότι υπάρχει πρόβλημα χρόνου. Όσοι επίκονται μπορούν να φύγουν. Εμείς θα περάσουμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξης, στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου. Επειδή είναι και κλεισμένο το θηρόν αυτό το τμήμα της συνεδρίασης, παρακαλώ όσοι δεν δικαιούνται να είναι μέσα, ας αποχωρήσουν από την αίθουσα. Και ενώ όσους δεν έχουν ε, την